Uh, so good uh, Καλό σας απόγευμα. Συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση. Ήμουν με το Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου για μια σύντομη συνάντηση. Αλλά οι συζητήσεις ήταν ε, χρήσιμες για τα μέλη. Γιατί δεν εγκρίθηκε η αποστολή στο Δουβλίνο. Αυτό ήταν το θέμα. Καλώς ορίζω θερμά όλους στην απογευματινή συνεδρίαση. Για όσους δεν είσαστε εδώ το πρωί και όσοι τώρα μπαίνουν στο διαδίκτυο, έχουμε ένα καινούριο newsletter, έχει εκδοθεί, οπότε μπορείτε να το ψάξετε στο διαδίκτυο. Και δεύτερον, αν ε, σας αρέσει το Twitter, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς έχει τώρα και λογαριασμό στο Twitter, και ήδη η κυρία Στάιλερ έκανε twittering και έχουμε και σύμβολη από πολίτες όπως λέγαμε σήμερα το πρωί. Οπότε μπορεί να υπάρχουν ενθουσιώδεις πολίτες και για τις δημόσιες ε, συμβάσεις. Η διεύθυνση είναι EP, κάτωτε ε, παύλα, single, mm, mm, single market, όλο μαζί, EP, κάτω παύλα single market, το Twitter hashtag και όσοι ε, αρέσκονται στο Twitter, ο εισηγητής μας είναι, είμαι βέβαιος, μπορείτε να προσθέσετε λοιπόν και εσείς ένα link από το δικό σας Twitter site. Ε, ευχαριστώ κυρία Πραντεργάς. Εγώ δεν είμαι στο Twitter. Είναι μια πρόσφατη εφεύρεση που δεν με έφτασε ακόμα. Μπορεί, μπορεί να πιστώ. Ακόμα δεν έχω πιστεί όμως. Λοιπόν, αυτό ήταν σημαντική ανακοίνωση. Τώρα θα... Την επόμενη ώρα θα κάνουμε μια δημόσια συζήτηση για την κατάσταση πραγμάτων στην Οδηγία Δημόσιων Συμβάσεων και φαντάζομαι ότι θέλετε να ξέρετε την πρόοδο όλοι. Όλοι γνωρίζουν βέβαια, αλλά αρχίζω τη συζήτηση λέγοντας ότι μετά από λεπτομερή συζήτηση με όλους τους σκιώδεις και τους συντονιστές, αποφασίσαμε να αναβάλουμε την ψηφοφορία στην Επιτροπή γιατί μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου. Γιατί θεωρήσαμε ότι χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρώσουμε μια αναθεώρηση όλων των τροπολογιών σε βάθος και υπάρχει βέβαια και το θέμα των συμβιβαστικών που είναι πολύ σημαντικές. Θα υπάρξουν ε, πολλές ψηφοφορίες και στις συμβιβαστικές. Η ποιότητα της δουλειάς μας ε, γύρω από τις συμβιβαστικές, όπως σε κάθε πρόταση, επηρεάζει την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Και αυτό ήταν η απόφαση που προτάθηκε. Είναι σημαντικό να είναι ενήμεροι όλοι. Θα συζητήσουμε λοιπόν για μία ώρα σήμερα και αύριο το, όχι, αύριο το πρωί, από τις 9 μέχρι τις 10, δηλαδή η αυριανή συνάντηση, η συνεδρίασή μας, Λοιπόν, η συνεδρίαση 9 ε, με 10 και 45 αύριο θα είναι και κλεισμένων των θυρών και θα, είναι, θα προεδρεύει ο εισηγητής ε, για τις συμβιβαστικές τροπολογίες και στις 10 και 45 θα συναντηθεί σε πλήρη σύνθεση η Επιτροπή. Είναι σαφές. Αυτό και για όσους παρακολουθούν. Λοιπόν, μεγάλη μακροσκελής η εισαγωγή μου αυτή τη φορά. Τώρα θα δώσω τον εισηγητή στο, θα το λόγο στον εισηγητή τον κύριο Ταραμπέλα για να μας πει πώς έχουν τα πράγματα και θα βρείτε και συμβιβαστικές τροπολογίες 1 με 31 στα φάκελο έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Έτσι, το υπογραμμίζω αυτό γιατί δεν είναι οριστικές. Σας δίνουν όμως σαφείς ενδείξεις για το πού προς τα που πάνε τα πράγματα. Μάρκ Ταραμπέλα, έχει το λόγο λοιπόν για να παρουσιάσει το θέμα στην Επιτροπή της τροπολογία. Ε, Τροπολογίας. Οι σκιώδει θα σχολιάσουν, θα κάνουμε και μετά γενική συζήτηση. Και ε, χαίρομαι που καλωσορίζω τον Κλάου Βίντνερ και την ομάδα του, τη σκληρά εργαζόμενη ομάδα του από την Γενική Διεύθυνση αγορά και θα του δώσω το λόγο όταν έρθει η ώρα να μιλήσει για τα θέματα που θα έχουν τεθεί. Παρακολουθεί πολύ και το Συμβούλιο. Ε, κύριε Ταραμπέλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καταρχήν ευχαριστώ τους συντονιστές που κατάλαβαν τη σκοπιμότητα να μην ψηφίσουμε αύριο και να βάλουμε για 15 μέρες την ψηφοφορία, διότι λόγω των πολλών συνεδριάσεων που είχαμε, τεχνικές συνεδριάσεις και πρέπει να δούμε τις διαφορετικές. Να ευχαριστήσουμε ε, το προσωπικό των πολιτικών ομάδων και της Επιτροπής ΙΜΚΟ που δούλεψαν σκληρά και συνεπώς ήταν λογικό να ανασταλεί για λίγο χρονικό διάστημα η ψηφοφορία για να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς λαμβάνοντας υπόψη πολλού παράγοντε προ το συμφέρον όλων και προ το συμφέρον του Κοινοβουλίου, ώστε να υπάρχει μια κοινή τοποθέτηση. Διότι για τις δύο οδηγίε υπήρχαν 2.500 τροπολογίε και δεν πρέπει να είναι πολύ βαριά τα κείμενα, πρέπει να τα ελαφρύνουμε λίγο. Γι' αυτό κατά την άποψή μου ήταν απαραίτητο να δώσουμε ακόμα 15 μέρες χρόνο για να υπάρξουν συμβιβασμοί. Γνωρίζοντα, όπω είπατε πρόεδρε, ότι η ψηφοφορία προβλέπεται στις 18 Δεκεμβρίου την κλασική οδηγία, 24 ε, Ιανουαρίου 2013 για την τομεακή οδηγία και αύριο θα έχουμε μια συνεδρίαση πάνω σε σημαντικά clusters στρατηγική σημασία των δημοσίων συμβάσεων, το cluster 2, άρθρο 1, αλλά αύριο και στις 6 Δεκεμβρίου θα υπάρξει shadow meeting για τι τις τελευταίες ελπίζω λεπτομέρειες και του συμβασμού σε τομεακό επίπεδο. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε τα κλάστερ 1, 2, 4, 7, 8 και 9, δηλαδή την επιλογή των διαδικασιών, τις διαδικασίες συμβάσεων, procurements, την βελτίωση των διαδικασιών, τις άλλες διαδικασίες και την διακυβέρνηση. Συνεπώς σήμερα Νομίζω ότι φτάσαμε σε σχετικά καλό αποτέλεσμα για τα δύο πρώτα clusters που αναφέραμε, διότι αυτές οι θεματικές είναι λιγότερο εμφυλογόμενες μεταξύ μας. Και για τα κλάστερ 7 και 8, για να δούμε τις παραλλαγές, τις τροποποιήσεις των ε, ε, δημοσίων συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, νομίζω ότι καταλήξαμε σε καλούς συμβασμούς ισορροπημένου που εξασφαλίζουν είτε την ευελιξία που απαιτείται από τις ε, ε, δημοκρατικές αρχές και από τις επιχειρήσεις, είτε αρκετή διαφάνιση δικασίες κυρίως για το αντικείμενο ε, του άρθρου 18, εμπιστευτικότητα, άρθρο 21, σύγκρουση συμφερόντων. Λόγω της ευελιξίας που προβλέπεται πρώτα απ' όλα στην πρόταση Επιτροπής και το κλάστερ το οποίο εθελεί το Κοινοβούλιο, νομίζω ότι το κλάστερ 9 που αφορά τη διακυβέρνηση είναι πολύ σημαντικό, επειδή ε, συνιστά μια ισορροπία μεταξύ ευελιξίας για τις δημοκρατικές αρχές και την απαραίτητη χρηστή διακυβέρνηση που χρειάζεται με τη διαφάνεια και με σωστούς διοντολογικούς κανόνες που πρέπει να βελτιωθούν. Οι ασάφειες παραμένουν όσον αφορά την αρχή ελέγχου, στην οργάνωση των κρατικών εξουσιών, δηλαδή σε ποιο επίπεδο ε, τα ομοσπονδιακά κράτη πρέπει να προσδιορίσουν ε, την εξουσία τους. Ε, επιδείξαμε ρεαλισμό, ε, λαμβάνοντα υπόψη το καταστάσιο σε διάφορα κράτη-μέλη και με αυτή τη συμβαστική λύση έχουμε μια πιο ελαφρά διαδικασία, εξασφαλίζοντας καλό επίπεδο ελέγχου στην Ευρώπη και σε ορισμένε χώρε υπάρχει ήδη αρκετό έλεγχο. Η διακυβέρνηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο λόγω ε, των περιθωρίων ελιγμών των διαπραγματεύσεων που έχει η Δημοκρατική Αρχή και γι' αυτό στην πρώτη μου έκθεση ε, ανέφερα ότι χρειάζεται μια αρχή ελέγχου στη χώρα, αλλά εκεί που υπάρχει μπορεί να δημιουργηθεί μια νέα αρχή ανάλογα με τις διαδικασίες που ισχύουν σε κάθε χώρα. Και αυτό αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 84. Προτού δώσω το λόγο στους συναδέλφους, θα ήθελα να σας πω ότι τα πιο σημαντικά θέματα και τα πιο ακαθόδη είναι εκείνα τα οποία μας διαφοροποιούν το περισσότερο και εκείνα θα φύγουν αύριο μεταξύ 9 και 11 παρατέταρτο και θα είναι πολύ πιο δύσκολο εκεί να επιτευχθεί συμφωνία επί ε, των προσφορών ε, ιδιαίτερα χαμηλών που μας προστατεύουν από κοινωνικό ντάμπινγκ κατά κάποιο τρόπο αλλά και τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των κοινωνικών κριτηρίων και το σκέλος της υπεργολαβίας άρθρο 71 κυρίως. Θα ήθελα να προσθέσω, δεν το είπα, σχετικά με το κλάστρο 8, το αποτέλεσμα είναι αρκετά καλό. Μίλησαμε πολύ για τις ε, δημοκρατικές αρχές. Είναι οι πρώτες οι οποίες πρέπει να αφομοιώσουν και να εφαρμόσουν τις οδηγίες ε, που εκπονούμε τώρα. Δεν λησμονήσαμε όμως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την καλύτερη πρόσβασή τους ε, στις δημόσιες συμβάσεις, στις ε, κρατικές προμήθειες στις οποίες συμμετέχουν λίγο σήμερα, κυρίως μέσω της συνενένωση πολλών μικρών επιχειρήσεων, ώστε να διευκολυθούν οι καλές πρακτικές και αυτό ήταν ένα από τα light motive, αν θέλετε, τα οποία επανέλαβαν όλοι σχεδόν οι συνάδελφοι, δηλαδή να επιτρέψει, όπως και η αρχική οδηγία της Επιτροπής, που έλεγε ότι παρά τις δυσκολίες μας, ε, κατορθώσαμε να συμφωνήσουμε πάνω σε ορισμένε έννοιες, Παρόλο που θα καταλήξουμε ελπίζω σε κάποια συμφωνία, είχαμε την τύχη όμως ότι βασιστήκαμε σε μια πρόταση της Επιτροπής που ακολουθούσε την καλή κατεύθυνση. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, γιατί δεν συμβαίνει πάντοτε. Και μας επέτρεψε αυτό από την αρχή να ξεκινήσουμε με μια καλή βάση, υπογραμμίζοντας το γεγονός ε, συνάντησα χθε την Προεδρία, τη Μελλοντική Προεδρία της Ιρλανδίας με την προηγούμενη, την πρέσκο, σχεδόν προηγούμενη, την ε, Προεδρία της Κύπρου που τελειώνει τώρα και μαζί τους συζήτησα ότι πρέπει να έχουμε την ίδια μέθοδο εργασία και ελπίζω ότι στο μέλλον θα μπορούμε με ευκολία να συγκρίνουμε τις συμφωνίες και τις διαφωνίες μας επάνω στα διάφορα κλάστερ. Αυτή είναι η μέθοδος την οποία εισήγαγε η Προεδρία της Δανίας και την χαιρετίζουμε. Τώρα ακούω τις παρατηρήσεις σας, τις κριτικές σας, αλλά και τα χειροκροτήματά σας αν υπάρχουν. Oh, well, I'm sure some words of praise. Um, so, um, uh, so let's, let's see. Um... Βέβαια υπάρχουν παρατηρήσεις. Θα έλεγα γενικά ότι εάν δούμε τη δουλειά που έγινε, κοιτάζοντας τα όσα έγιναν για το συμβιβασμό και τις τροπολογίες ε, που αντικαταστάθηκαν από ε, συμβιβασμού, θα δείτε ότι έγινε μεγάλη πρόοδος. Ε, ευχαρίστησε, πρέπει να ευχαριστήσουμε και το προσωπικό μας βεβαίω και τον εισηγητή, αλλά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε πολλούς τομείς. Κοιτάζοντας λοιπόν τις τροποποιήσεις για μακρόν καταλήξαμε στο ότι το αρχικό σας κείμενο ήταν το καλύτερο. Κατά την άποψή μου λοιπόν, η διαδικασία υπήρξε καλή, διότι δοκιμάσαμε, αν θέλετε, το έγγραφο της Κομισιόν σε σχέση με τις προτάσεις βελτίωσης που έκαναν οι συνάδελφοι. Και καταλήξαμε ότι το έγγραφο της Επιτροπής ήταν το καλύτερο. Πρέπει αυτό να μας ενθαρρύνει. Συνοψίζοντας λοιπόν, υπάρχουν καλά πράγματα εδώ και αυτό είναι το πνεύμα που θα μας καθοδηγεί. Ο κύριος Σάγκλη δεν είναι εδώ, ο κύριος Φάρ θέλει να μιλήσει εξ ονόματός του. Νομίζω ότι είναι στο Σουρινάμ, δεν απατώμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιστρέφει τώρα. Αλλά μου ζήτησε να κάνω ορισμένα σχόλια εξ ονοματός του. Θα έρθει αργότερα εδώ. Αλλά θέλω να σας πω, αγαπητέ κύριε Σιγητά, ότι για τα χειροκροτήματα δυστυχώς εμείς δεν βρήκαμε λόγους, αλλά θα είμαστε πολύ ευγενείς και μαλακοί σήμερα, διότι πιστεύουμε ότι η προτινόμενη αναβολή είναι κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει ώστε να βρούμε σοβαρούς συμβιβασμούς. Όπως... Σε αυτές τις ομάδες τώρα 1, 4, 7, 8, 9 θα πω κάποια πράγματα. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Καταρχήν να πω, επειδή επενέσατε την Κομισιόν, ότι κατά τη γνώμη μου, και δεν το λέω ε, όν εκ των υστέρων προφήτης, αλλά νομίζω ότι πάμε στην τελική ευθεία με τις διαβουλεύσεις. Αρχίζουν να διαφαίνονται καλές συμβιβαστικέ τροπολογίες, αλλά σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες που δεν ε, δημιούργησα εγώ, οι προσδοκίες ότι θα απλουστευτεί το σύστημα, αυτό δεν υλοποιήθηκε. Ίσως ε, και η Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει απλούστερη, μπορεί να μην γίνεται, αλλά νομίζω ότι είναι τελείως λάθος να δημιουργούμε την εντύπωση ότι απλοποιήθηκε. Νομίζω ότι σε ορισμένα σημεία δυσκολεύουν μάλιστα και λίγο τα πράγματα και γι' αυτό ήμουν ε, λίγο επιφυλακτικός αν χρειάζεται αυτή η επεξεργασία. Τώρα πάντως πρέπει να κάνουμε το καλύτερο αφού υπάρχει. Λοιπόν, ε, σε σχέση με τον, το τι λέει ο κύριος Έγγελος Κιώδης μας για τις ομάδες. Καταρχήν καλό είναι που βρήκαμε τη συμβιβαστική λύση όλες οι διαδικασίες για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων να πρέπει να ε, ε, ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο. Έτσι υπάρχει η δίκαιη δυνατότητα ο εθνικός νομοθέτης να μπορεί να εφαρμόζει στις εθνικές διατάξεις όλα αυτά που αποφασίσαμε. Επίσης για τις προθεσμίες ε, αυτές ανταποκρίνονται περίπου στις αρχικές προτάσεις της Κομισιόν και αυτές τις βλέπουμε πολύ θετικά και χαιρόμεθα επίσης ε, διότι ε, δημιουργούνται και προτάσεις ε, για τις συμπράξεις καινοτομία. Αυτό είναι καλό ότι ενσωματώθηκε και μπορεί να συγκεντρώσει την πλειοψηφία στην ομάδα που συζητούμε. Τώρα, η ηλεκτρονική ανάθεση μετά από δύο χρόνια από τη θέση σε ισχύ θα ε, διατίθεται για όλους. Σε κάποια κράτη-μέλη θα υπάρξουν κάποιες δυσκολίες ε, στην ε, μετάβαση, αλλά γενικά νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε διαφανείς στην εσωτερική αγορά, παρόλο που θα υπάρξουν κάποιες αναπροσαρμογές δύσκολες σε κάποια κράτη-μέλη. Να πω σε αυτό το σημείο ότι το procurement passport, αυτό το ενιαίο έγγραφο διαβατήριο, πώς να το πούμε, ε, θα έρθει και ο, έρχεται και ο Σκιώδης, δεν ξέρω πώς το λένε στα γερμανικά, διαβατήριο ε, συμβάσεων. Ε, φαίνεται ότι στο Συμβούλιο απομακρύνθηκε, δεν υπάρχει πια. Αυτό και για μας και για το ΕΛΚ ήταν σημαντικό ούτως ώστε οι ΜΜΕ να συμμετέχουν στη διαδικασία των αναθέσεων. Γι' αυτό θα ήθελα να μην αφήσουμε το Συμβούλιο να το βγάλει αυτό το στοιχείο του διαβατηρίου από το κείμενο και θα πρέπει να έχει και τουλάχιστον ενός έτους διάρκεια το διαβατήριο αυτό για δεν ωφελεί. Για τη διακυβέρνηση, το governance, βελτιωμένη εποπτεία για την Κομισιόν για το πώς εφαρμόζεται το δίκαιο αναθέσεων σε επίπεδο κρατών μελών. Νομίζω ότι πρέπει να δεχτούμε ότι το Συμβούλιο θα επιβάλλει τη συμβιβαστική λύση που, ε, στην οποία κατέληξαν. Δεν κακή συμβιβαστική λύση, γιατί και εγώ, ε, ως εισηγητής για την ε, ενιαία διακυβέρνηση στην εσωτερική αγορά, ε, αυτό μας διευκολύνει γιατί η εφαρμογή θα ε, επιτρέπει καλύτερη εποπτεία του συστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, έτσι είμαστε αρκετά κοντά και γι' αυτό άλλωστε μπορέσαμε να βρούμε και ικανοποιητικέ συμβιβαστικέ τροπολογίες. Ευχαριστώ. Σα Frank, welcome. Did you, um, did you wish to Σας, ευχαριστώ. Ε, καλώς Φρανκ. Θέλεις να προσθέσεις κάτι στα όσα είπε ο συνάδελφος. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Προς το παρόν θα σταθώ σε αυτά που είπε ο συντονιστής μου. Ε, είμαι λίγο συγχυσμένος, θέλω ένα-δυο λεπτά να συνέλθω και μετά μπορεί και να επανέλθω. Ωραία. Ποιος έχει σειρά. Ο κύριος Κρόιτσμαν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ και εγώ. Αυτό ήταν Ηράκλειο έργο και για τη γραμματεία και για τον εισηγητή. Καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι περιπλέκουμε μάλλον τα πράγματα και υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι η Κομισιόν έχει κάνει μια ισορροπημένη, πολύ ισορροπημένη πρόταση και θα πρέπει να κάνουμε λίγο πίσω στις ε, απαιτήσει μας. Παράκληση επίσης να είμαστε πιο ευέλικτοι σε ό,τι αφορά τις διάφορες προτάσεις. Τώρα έχουμε τις ομάδες 1 με 4, συμφωνούμε, τις υποστηρίζουμε, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς πρέπει να πούμε ότι έχουμε εράκλειο έργο και μπροστά μας, γιατί τα επίμαχα θέματα θα τα δούμε αργότερα. Καλό είναι να εισαχθεί γρήγορα το ηλεκτρονικό σύστημα γιατί έτσι ε, εξοικονομούνται κάποιες δαπάνες και το διαβατήριο, όπως είπε ο συνάδελφος Σβάμπ, φαίνεται καλό. Από ό,τι φαίνεται το Συμβούλιο δεν το θέλει. Ε, Επίση, ε, το σύστημα IMI, το σύστημα πληροφόρηση για την εσωτερική αγορά, πρέπει να το ενεργοποιήσουμε. Δεν έχουμε αντίρρηση, αφού υπάρχει, γιατί να μην το αξιοποιούμε και αυτό το IMI φαίνεται να ε, δίνει κάποια πλέον εκτίματα. Παρ' όλα αυτά, το διαβατήριο, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, θα διευκολύνει τις διαδικασίες και προφανώς ε, αν εκδώσω διαβατήριο για ένα χρόνο και εντωμεταξύ ε, διαπραχθεί αξιόπινη πράξη, βεβαίως θα υπάρξει αλλαγή αυτό θα είναι μια ατυχία, αλλά το ίδιο θα συνέβαινε αν εξεδίδωτο για έξι μήνες και μετά υπήρχε πρόβλημα. Εμείς το υποστηρίζουμε, συνάδελφε Σουάρτ. Στην επτά ομάδα θέλουμε αν υπάρχουν εναλλακτικέ προσφορές να ε, ε, δικαιολογούνται. Και στο 8 υπάρχουν πολλές ορθές διαδικασίες, αλλά χρειάζονται βελτιώσεις. Ε, τώρα, η προστασία στην αιτιολογική σκέψη αυτών που αποκαλύπτουν προβλήματα, δεν υπάρχουν παντού συμβούλια επιχειρήσεων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Ε, άρα αυτό το μέσο μπορεί να έχει νόημα. Σε περιπτώσει συγκρούσεων ε, συμφερόντων συμφωνούμε με τον εισηγητή ε, που προσανατολίζεται στο απλούστερο κείμενο του Συμβουλίου. Γενικά η διαδικασία είναι θετική, αλλά στο 39.1 ε, νομίζω ότι ε, η διαγραφή των διαβουλεύσεων δεν είναι καλή. Για την ε, τροποποίηση η αλλαγή των συμβάσεων ε, έχουμε στο 72.35 μια τροπολογία. Στο 9 μπορούμε να συμφωνήσουμε με πολλά. Κάποια χρήζουν διαπραγματεύσεων υπέρ της διαγραφής του 84 εθνική εποπτεία με βάση το άρθρο 83. Επίσης είπαμε ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υπάρχει βοήθεια ε, όταν εφαρμόζονται οι διατάξεις ε, ανάθεσης. Είμαστε κατά του 85 ε, για θα πρέπει εδώ να υπάρχουν για τους υπεργολάβους. Α, εδώ προβλέπεται ενημέρωση για τους παροχή πληροφοριών για τους υπεργολάβους. Αυτό είναι πολύ γραφειοκρατικό. Εμείς είμαστε υπέρ της απλοποίησης και στην υποχρέωση υποβολής εθνικών εκθέσεων. Σταματώ εδώ και νομίζω ότι ακόμα έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε. Ε, έχει νόημα να, γι' αυτό ε, ότι αποφασίσαμε να αναβάλουμε λίγο την, ε, για λίγες εβδομάδες την ψηφοφορία γιατί νομίζω ότι εδώ πρέπει να δουλέψουμε σωστά ε, δεν είναι τόσο σημαντικό να δουλέψουμε γρήγορα όσο να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ όλους πολύ και ελπίζω ότι η μέχρι τούδε επικοδομητική συνεργασία μας θα συνεχιστεί και στις καυτές διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρούλη. Και εγώ να ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία μέχρι τώρα. Συμφωνώ με τον κύριο Σουάμπ και να του δώσω εκ των υστέρων δίκιο. Γιατί η πορεία των διαπραγματεύσεων με ε, προσγείωσε λίγο εις ό,τι αφορά τη δυνατότητα απλοποίησης. Φαίνεται ότι... Ε, αν πηγαίναμε προς τη, τον κανονισμό, ίσως θα ήταν διαφορετικά. Ε, είναι λίγο πιο μπερδεμένο το θέμα της οδηγίας. Γι' αυτό ε, η... και επίσης η πρόταση της Κομισιόν είχε μπήκε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Πώς να γίνει η απλοποίηση. Η μόνη απλοποίηση από αυτή την οδηγία είναι η ηλεκτρονική ανάθεση όταν θα μπορεί να υπάρχει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα δώσει όθηση σε μεγαλύτερη ασφάλεια και απλοποίηση, αλλά είναι το μοναδικό που μπορούμε να πούμε προς αυτή την κατεύθυνση, ότι θα απλοποιηθεί δηλαδή. Κατά τα άλλα, συμφωνώ με την ανάλυση του κυρίου Schwab, ε, το toolbox, ε, η εργαλειοθήκη αυτή είναι χρήσιμη, δεν υπήρχε μέχρι τώρα σε όλα τα κράτη-μέλη και είναι καλό ότι θα υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη και το θέμα των προθεσμιών είναι ικανοποιητικό ως προς τη ρύθμισή του. Για το διαβατήριο εξανάθεση έχω κάποια προβλήματα γιατί προσωπικά μου φαίνεται ότι είναι δυσκίνητο, είναι πολύ μακρά διαδικασία. Θα προτιμούσα να είναι πιο απλό το κείμενο ε, και να ξέρουμε τι θα πρέπει να καλύπτει αυτό το διαβατήριο προβλέπει πάρα πολλά μπορεί να είναι πιο απλό για να ε, ωφελήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό δεν έχουμε προσυπογράψει τη συμβιβαστική ακόμα. Τώρα, θα αναφέρω και δύο-τρία άλλα πράγματα ε, σε σχέση με την ομάδα 2. Εκεί πιστεύω ότι το κείμενο ε, της τροπολογίας 13 που αναφέρεται στο άρθρο 15 δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που συζητήσαμε στη συνάντηση των σκιωδών και θα ήθελα αύριο να το διευκρινίσουμε αυτό το θέμα γιατί το κείμενο είναι διαφορετικό από εκείνο που είχα σημειώσει εγώ ως συμβιβαστική τροπολογία την τελευταία φορά, την περασμένη φορά. Ε, το λέω και προς τον εισηγητή, γιατί νομίζω ότι και εκείνος θεωρούσε σημαντικό το άρθρο 15. Οπότε να ελέγξουμε αν όντως ήταν αυτό το συμβιβαστικό κείμενο. Επίσης, θέλω να συζητηθεί στις ομάδες 8 και 9. Εδώ πρόκειται για μικρολεπτομέρειες, αλλά προσωπικά θεωρώ ότι, για παράδειγμα, το άρθρο 86 μπορούμε να το, και να το διαγράψουμε. Θα ψηφίσουμε. Εκεί ε, δεν θα συμμετάσχουμε στη διοπολογία δηλαδή. Και πρέπει να το διευκρινίσουμε, γιατί εγώ είχα καταλάβει ότι η τροπολογία 21 στο άρθρο 16 δεν περιλαμβάνει το εδάφιο για τα κονσόρτσια το, ε, αυτό αναφερόταν στην αιτιολογική σκέψη. Τώρα έχουμε και την τροπολογία και την αιτιολογική σκέψη. Θα το ρυθμίσουμε και αυτό στην αυριανή συζήτηση. Πάντως δουλέψαμε καλά και νομίζω ότι και στις άλλες ομάδες θα προχωρήσουμε γρήγορα. Um, just, uh, this is my, uh, θα μιλήσω λοιπόν με τον ρόλο μου ως και ο και ε, παρεμπιπτόντως οποιοδήποτε άλλο θέλει να συνεισφέρει στη συζήτηση μπορεί κάλλιστα να το κάνει εννοείται. Ε, κάντε μου ένα νόημα, όποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο για την συγκεκριμένη πρόταση. Καταρχάς λοιπόν να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα διότι θεωρώ ότι καταλήξαμε σε καλή συμφωνία καταρχάς ε, για τις ε, συμπράξεις καινοτομία, που είναι ένα νέο εργαλείο για τις δημόσιες συμβάσεις και να περάσω στο θέμα της απλοποίησης στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Βάμπ. Το να προσθέσουμε και νέα μέσα μπορεί να κάνει πιο μακροσκελή την ε, νομοθεσία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα περιπλέξει απαραίτητα και την εφαρμογή της. Το να έχουμε μία ε, σύμπραξη καινοτομία είναι τελείως διαφορετικός τρόπος ε, ανάθεσης. Ε, και θα είναι πολύ σημαντικό και για τους πελάτες και για τους προμηθευτές. Θα δημιουργήσει νέες σχέσεις, ε, θα βελτιώσει την ποιότητα του αποτελέσματος και όσον αφορά το κόστος ε, και όσον αφορά την τεχνολογία. Και υπάρχουν και άλλες σημαντικές πτυχές, όπως για παράδειγμα βιωσιμότητα, κατάλληλη χρήση ενέργειας και κατάλληλη χρήση για τους χρήστες, για τους πελάτες. Για όλους αυτούς λοιπόν τους τομείς θεωρώ ότι το βασικό βασικό στοιχείο της απλοποίησης είναι ουσιαστικά η ποιότητα της ίδιας της διατύπωσης και το κατά πόσο είναι επίκαιρη η νομοθεσία μας. Και σε αυτά τα θέματα χρειάστηκε να ε, αντιμετωπίσουμε με τους κανονισμούς όσοι έχουν αυτή τη στιγμή. Και εδώ τίθεται και το ζήτημα. Εάν δώσουμε αυτό στον κόσμο, θα πρέπει να διαπιστώσουν ότι πρόκειται για βελτίωση, διότι είναι πολύ πιο σαφές, καταλαβαίνουμε τι πρέπει να κάνουμε, οι προσυμβατικές διαδικασίες είναι πολύ πιο απλές ε, και ως αναθέτουσα αρχή έχουμε πολλά εργαλεία στη διάθεσή μας. Ε, υπάρχει μεγαλύτερο πεδίο διαπραγμάτευσης που ελπίζουμε ότι θα μας οδηγήσει και σε καλύτερα αποτελέσματα, κάτι το οποίο επιτυγχάνουμε χωρίς να μειώσουμε και την ανταγωνιστική φύση της αγοράς. Και αυτό θεωρώ ότι βοηθάει ιδιαίτερα και το κόστος της διακυβέρνησης, διότι νομίζω ότι ήταν απόλυτα σαφέ ότι ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι ότι δεν εφαρμόζονται με μεγάλη συνέπεια οι κανόνες αυτή τη στιγμή. Και ένα από του λόγου που δεν εφαρμόζονται όπω πρέπει είναι και γιατί είναι αρκετά δυσνόητοι. Και επειδή ακριβώ είναι τόσο δυσνόητοι, γνωρίζουμε ότι ο κόσμος προσπαθεί να βρει τρόπο να τα παρακάμψει. Εάν όμω είναι πολύ πιο φιλική προς το χρήστη οι κανόνες, καταρχάς ε, ε, θα ε, είναι ανασταλτικό παράγοντα αυτό για όσους θέλουν να κάνουν κατάχρηση και επίσης θα υπάρχουν και βελτιώσεις. Επίσης, ε, χρειαζόμαστε και ένα μηχανισμό παρακολούθησης και νομίζω ότι είναι ε, αποδεκτό από όλου ότι ο μηχανισμός που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν απόλυτα σωστός, διότι υπήρχαν αρκετές χώρες που είχαν αρκετά καλά ε, συστήματα και μπορούσαν να κάνουν τον έλεγχο όπως πρέπει. Και, και πάλι να πω εδώ ότι ο τρόπος που θα το διατυπώσουμε ε, θα μας οδηγήσει σε μια προσέγγιση που μας ενδιαφέρει κυρίως το αποτέλεσμα. Θα υπάρχει ένα θεσμικό οργανισμό που θα παρακολουθεί τις δημόσιες συμβάσεις, που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν εξαρτάται πώ θα μα τα δώσουν, αλλά αυτά απαιτούνται. Πρέπει να υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Και το τι θα έχουμε ως αποτέλεσμα από το σύστημα είναι αυτό το οποίο πρέπει να εξετάσουμε κατά βάση. Ε, όσον αφορά τώρα τις τροπολογίες, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε καταφέρει να ε, κάνουμε τόση πρόοδο. Και οι σημαντικές ομάδες τροπολογιών για τα στρατηγικά σημεία ε, είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε δεν είμαι βέβαιος κατά πόσο θα έχουμε συμβιβαστικέ προτάσεις ε, για τα πάντα. Κάποια πρέπει να τα ψηφίσουμε. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε και τις ψηφοφορίες, αρκεί βέβαια ε, να τηρήσουν όλο το αποτέλεσμα στη συνέχεια και να μπορέσουμε να το προασπίσουμε στις μελλοντικέ διαπραγματεύσει. Αυτά λοιπόν είναι σημαντικά και γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε και περισσότερο χρόνο να τα συζητήσουμε και θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και λίγο το χρόνο μας για να δούμε λίγο τι γίνεται με τις τροπολογίες. Υπάρχουν κάποιες διατυπώσεις που είναι μάλλον περιτές, δεν προσθέτουν τίποτα στο χαρακτήρα του κειμένου. Για παράδειγμα, για για τις εναλλακτικέ προσφορές νομίζω ότι συμφωνήσαμε ότι πρέπει να επανέλθουμε στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς ε, θα χρησιμοποιείται αυτή η νομοθεσία για να μπορέσουμε να κάνουμε μια τελική ε, αναδιατύπωση και να φροντίσουμε όταν θα έχουμε το κείμενο και θα είναι δημόσιο ε, να υπάρχουν κάποιες καλές ιδέες ε, και ελπίζω αυτές να τις έχουμε τις επόμενες εβδομάδες γιατί είναι πολλές ενδιαφέρουσες οι ιδέες αυτές οι οποίες θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε το κείμενο. Σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένο. θα συνεχίσω να συμμετέχω ενεργά και ως σκιώδης εισηγητής αλλά και ως πρόεδρος της Επιτροπής και τώρα ξαναλαμβάνω τα ενία ως πρόεδρος και να σας πω ότι αύριο το πρωί στην συνεδρίαση που θα γίνει για τα πρώτα τρία τέταρτα θα κάνουμε μια κοινή συνεδρίαση με τον κύριο Ζουβά και τον κύριο Ταραμπέλα για να συζητήσουμε τα διαφιλονικούμενα ζητήματα για την οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις και την οδηγία για τις παραχωρήσεις. Και θα υπάρξει και συζήτηση για τις παραχωρήσεις ε, αργότερα, τις συμβάσεις παραχώρησης. Νομίζω ότι καταφέρνουμε σιγά σιγά να έχουμε όλο το κείμενο για τις δημόσιες συμβάσεις που είναι πολύ ε, θετικό κατά την απόψή μου. Να σας υπενθυμίσω βέβαια ότι υπάρχουν κάποια θέματα ορίων μεταξύ των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης τα οποία πρέπει να θέσουμε. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο το λόγο. Εγώ, κύριε Διόγκ, ζητώ συγγνώμη, ε, δεν σηκωθήκα τόρτες για να σας δω. Έχετε το λόγο. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Ο κύριο Σαλβίνη λείπει. Ο κύριο Μπαλτασάρε θα λάβει το λόγο μετά. Κάποιο άλλο. Άλλοι συνάδελφοι. Και ο κύριο Έγκελ θα μιλήσει. Ο κύριο Διόν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, συμφωνώ με το έργο του εισηγητή που είναι εξαιρετικό. Να αναφέρω κι εγώ κάποια πράγματα. Το άρθρο 15. Εδώ η συμβιβαστική νομίζω είναι πολύ καλή. Και έχω ένα πρόβλημα δεν καταλαβαίνω γιατί είναι συμβιβαστική. Αυτή αφορά το άρθρο 21, ε, σύγκρουση συμφερόντων. Γιατί ξαναγυρίζουμε σε τόσο γενική διάταξη. Η Διεθνής Διαφάνεια έχει καταθέσει μια έκθεση που λέει ότι συχνά γίνονται λάθη στις δημόσιες συμβάσεις και υπάρχουν συγκρούσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Γι' αυτό ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα Αυτό που δίνουν τις πληροφορίες για τις λειτουργίες, τους λεγόμενους whistleblowers, πρέπει να μπει στο προήμιο. Αλλά η κατάργηση των διατάξεων για τη σύγκρουση συμφερόντων θα είναι κρίμα. Τέλος, θα ψηφίσουμε στις 18 Δεκεμβρίου, είπαμε, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει αρκετός χρόνος για να έχουμε αξιολόγηση αμέσως μετά την ψηφοφορία σχετικά με το αν πρόκειται όντως για απλοποίηση. Εγώ το ζήτησα αυτό. Οι συνάδελφοι Σουάμπ και Ρούλε νομίζω ότι θα συμφωνήσουν ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, κάτι άλλο πολύ σημαντικό επίσης για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, μην μας ξεφύγει, γιατί το σύστημα πρέπει να ισχύσει και για τις ΜΜΕ. Να δούμε λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για να ε, πούμε εάν το κείμενο ανταποκρίνεται στα, σε αυτά που θέλουμε, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε στη συζήτηση για τα θέματα αυτά. Ο κύριος Παλτεσάρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον εισηγητή διότι κατάφερε να βρει μία λύση ε, την οποία συμμεριζόμαστε σε μεγάλο βαθμό για τα κλάστερ που συζητάμε σήμερα, τις ομάδες αυτές. Ε, να υπενθυμίσουμε ότι οι συμβαστικές προστάσεις στις οποίες καταλήξαμε είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικέ. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στις ομάδες 2 και 8, τις οποίες θα συζητήσουμε αύριο το πρωί, δεδομένου ότι εγώ δεν θα μπορέσω να συμμετάσχω, διότι ε, στην Ιταλία έχουμε κάτι μικρό προβληματάκια, ας το θέσω έτσι και πρέπει να επιστρέψω. Πρέπει όμως να θίξω κάποια ε, πράγματα. Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι πολύ συχνά ανακοινούμε τη σημαία της εσωτερικής αγοράς υποτίθεται για τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό και θεωρούμε ότι αυτά είναι θεμελιώδη προκειμένου να αναπτύξουμε μεγαλύτερη ολοκλήρωση στην Ευρώπη προ όφελο ε, του συστήματος των επιχειρήσεων μας, ε, των πολιτών μας και μετά όταν πρέπει να κάνουμε μια πιο θαραλέα χειρονομία αρχίζουμε όλοι να πιστοχωρούμε δεν λέμε ότι δεν θα έχουμε πια οδηγία, να κάνουμε κανονισμό, δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικά, να είναι όλα προαιρετικά, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι σε όλες τις οδηγίες στις οποίες ε, δώσαμε μάχη, αφήνοντας τις αρμοδιότητες ε, σε άλλους και περιμένοντας να κάνουν διάφορα πράγματα ε, λόγω καλής θελήσεως, τελικώς δεν είχαμε αποτελέσματα είχε μια προηγούμενη οδηγία που άφηνε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να ζητήσουν ε, αποζημίωση για τις ε, καθυστερήσεις ε, της δημόσιας διοίκησης. Επειδή όμως το αφήσαμε στα κράτη-μέλη να επιλύσουν το πρόβλημα, τελικώς δεν επιλύθηκε ποτέ το πρόβλημα. Και επομένως υποχρεωθήκαμε να κάνουμε οδηγία. Εγώ, αντίθετα, φρονώ ότι ακριβώς προκειμένου να ευνοήσουμε τη μεγαλύτερη ολοκλήρωση, είναι απαραίτητο όχι μόνο να ρυθμίσουμε κάποιες σημαντικές πτυχές της οικονομίας μας για τις δημόσιες συμβάσεις μας, αλλά να προσπαθήσουμε να έχουμε και μια πιο ομοιόμορφη νομοθεσία. Δεν μπορούμε να έχουμε μια οδηγία η οποία θα είναι διάσπαρτη με προαιρετικά στοιχεία και θα τα αφήνουμε όλα στα κράτη-μέλη και θα επιφύεται σε αυτά αν θα εφαρμόσουν το μεν ή το δε. Υπάρχουν κάποια στοιχεία της οδηγίας που πρέπει να είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Γι' αυτό λοιπόν για τα στοιχεία τα οποία με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, τις ομάδες 2 και 8 δηλαδή, τα οποία θα συζητηθούν αύριο, και πιο συγκεκριμένα τα άρθρα 71 και 69, καθώς επίσης και το 84, θεωρώ ότι όσον αφορά τις υπεργολαβίες είναι απόλυτα λογική η θέση να είμαστε υποχρεωμένοι να υποδεικνύουμε το ποσοστό της υπεργολαβίας ε, το οποίο ανατίθεται, όπως επίσης και στη δεύτερο παράγραφο είναι απολύτως απαραίτητο να προβλέπεται η δυνατότητα για την αναθέτουσα αρχή να πληρώνει απευθείας τον υπεργολάβο. αφήνοντας έτσι το ενδεχόμενο για μεγαλύτερη προστασία ε, του υπεργολάβου, ο οποίος δεν θα είναι στο έλεος του βασικού εργολάβου. Και αυτό δεν θα πρέπει να είναι προβλέπεται ή δεν προβλέπεται, γιατί ουσιαστικά αλλάζει την όλη διαδικασία. Και δεν θεωρώ ότι θα πρέπει... Ε, κάθε φορά σε κάθε κράτος μέλος να εφαρμόζεται κάτι διαφορετικό. Μια δεύτερη πτυχή. Άρθρο 69. Και εδώ θεωρώ ότι αποτείουμε φόρο τιμή στη διαφάνεια. Και δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε πίσω από γραφειοκρατικό άχθος που δεν υπάρχει στην ουσία. Εάν κάποιο ως ε, ε, διευθυντή μια επιχείρηση συμμετέχει σε ένα μειοδοτικό διαγωνισμό, τον οποίο κερδίζει μια άλλη επιχείρηση που κάνει μια προσφορά 30% χαμηλότερη από του υπολείπους γιατί ε, του ανατέθηκε ο διαγωνισμός ή θα τα αφήσουμε στη διακριτική ευχέρεια της δημόσιας διαίκησης να αποφασίσει αν θα μας ε, αιτιολογήσει γιατί του δόθηκε ο διαγωνισμός ή όχι. Αν λοιπόν υπάρχει ένα τέτοιο άρθρο, χωρί ποσοστά, 30, 40, 50, μετά θα καθορίσουμε ποιο θα είναι το ποσοστό, το οποίο δεν θέτει ένα όριο. Και δεν λέει ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και να είμαστε σωστοί προς αυτούς που συμμετέχουν στο μειοδοτικό διαγωνισμό. Και επομένω και μια άμεση και έμεση υποχρέωση της δημόσιας διοίκησης να δρά με διάφανο τρόπο και ε, δεν θα πρέπει να το αφήνουμε αυτό στην καλή θέληση των δημοσίων αρχών. Γιατί δεν θεωρώ ότι μετά από όλα τα αποτελέσματα και τι αναλύσει που απορρέουν για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι και πρωταγωνιστέ τη διαφάνεια. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι όσοι θέλουν να απορριθμίσουν αυτό το άρθρο και να μην υπάρχει καμία ρύθμιση να τα αφήνουμε στη διακριτική εκφέρεια των ε, δημοσίων διοικήσεων, κατά την άποψή μου λάθος κάνουν, διότι δεν βοηθούν αυτούς που θέλουμε να βοηθήσουμε δεν πιστεύω πραγματικά ότι είναι υπογραφειοκρατική υποχρέωση και ε, παρακολεί την απλούστευση μιας διαδικασίας το να μπορεί μια επιχειρήση να ζητήσει εξηγήσει γιατί κάποιος έχει κάνει πάρα πολύ χαμηλή προσφορά ε, μετά επιχείρηση που μπορεί η επιχείρηση, για παράδειγμα, που κέρδισε το διαγωνισμό να κατασκευάσει απευθεία τι πρώτε τα υλικά, επομένω ε, θα μπορέσει να ε, κερδίσει από εκεί. Ή θα κάνει κάποιε τεχνικέ βελτιώσει που θα τι επιτρέπει να έχουν τόσο φτηνή προσφορά. Αλλά δεν ε, θα μπορούμε να ελέγξουμε αν υποχρεώνουμε τους εργαζόμενους να δουλεύουν για παράδειγμα ώρες πολύ περισσότερες από όσες επιτρέπεται ή δεν πληρώνονται αρκετά. Μια επιχείρηση που κάνει πάρα πολύ χαμηλή προσφορά μπορεί μετά από ένα χρόνο, μετά από κάποιους μήνες που θα έχουν ξεκινήσει εργασίες, να δηλώσει ότι δεν είναι πλέον σε θέση να τηρήσει ε, τις δεσμεύσεις που ανέλαβε και ότι έχει ανέβει το κόστος για κάποιο υλικό π.χ. και να ζητήσει να συμπεριληφθεί και το υπόλοιπο 30%. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η θέση είναι απόλυτα λογική και γι' αυτό, και με αυτό ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι απόλυτα λογικό και το, αυτό που λέει ο εισηγητής για, την, ε, για τον έλεγχο. Όπου υπάρχουν δυνατότητες θα πρέπει να βρούμε μια λογική λύση διότι δεν θα πρέπει να είναι άλλη η αρχή που αποφασίζει. Εάν όμως δεν υπάρχουν, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος υπεύθυνο για τον διαγωνισμό, κάποιος τον οποίο μπορούμε να κάνουμε έκκληση αυτή τη στιγμή τεθεί σε εφαρμογή αυτή η οδηγία όταν θα την εγκρίνουμε, για να αμφισβητήσουμε το κατά πόσον ε, δεν εφαρμόστηκαν όλα όσα προβλέπονται από την οδηγία. Και πρέπει να υπάρχει αυτό. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θα πρέπει να ε, ε, απευθυνόμαστε απευθεία στις δικαστικέ αρχέ και να έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα οι δικαστικέ αρχέ. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι κάποιες ε, διαδικασίες, ιδίω αστικέ, πριν ξεκινήσουν έχουν μια καθυστέρηση 6-8 μηνών και μπορεί να πάρει και χρόνια η τελεσίδικη απόφαση. Επομένω θα πρέπει οι επιχειρήσει να μπορούν να απευθύνονται απευθεία στην αναθέτηση αρχή και δεν πρέπει να υποχρεώνονται να πάνε στη δικαστική αρχή. Αν του λέμε ότι δεν υπάρχει αρμόδια αρχή, τι θα λέμε ότι θα του τους προστατέσουμε τα δικαιώματά του 6 με 8 μήνε αργότερα και ότι δεν υπάρχει κάποιο υπεύθυνο, μια αρχή υπεύθυνη για να εφαρμόσει του κανόνε που θα εγκρίνουμε. Εάν θέλουμε να κάνουμε μια οδηγία και θέλουμε να έχει αποτελέσματα, τότε πρέπει να κάνουμε λύσει. Εάν θέλουμε να έχουμε μια οδηγία την οποία θα τη γεμίσουμε ευθύ εξ αρχή με κενά, τότε δεν θα λειτουργεί. Και πραγματικά εγώ δεν είμαι συνηθισμένο να δουλεύω για το τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι κανένας δεν έχει την πρόθεση να δουλεύει για το τίποτα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων. Και όπως είπα πρωτήτερα, η ποιότητα ε, της εργασίας είναι πιο σημαντική με την ποσότητα της νομοθεσίας. Ε, θα δώσω το λόγο στην Κλασβίνα. Ο κ. Μάντερς θέλει επίσης να μιλήσει, ο κ. Σάγκλ. Σας παρακαλώ να είσαστε όσο πιο σύντομοι ώστε να το πιο σύντομη, γιατί έρχονται και, έρχονται και άλλοι συνάδελφοι για το επόμενο θέμα. Ε, thank you, Chair. I just want to add... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλά θέλω να προσθέσω το εξή. Ήμουν σκιώδη ηγητής ε, στην Επιτροπή ΕΝΔΙ για αυτό το θέμα και εκεί καταλήξαμε στη συμφωνία για ε, την καινοτομία ως ένα σημαντικό κριτήριο για τις δημόσιες συμβάσεις. Εκείνο το οποίο είπαμε ήταν ότι οι κυβερνήσεις, οι αρμόδιες αρχές θα έπρεπε να είναι ο πελάτης και η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι βιτρίνα για την καινοτομία στο μέλλον και όχι να προσπαθεί να βρίσκει διάφορες άλλες θυγατρικές επιχειρήσεις για καινοτομίες. Κατόπιν έγινε συζήτηση με τον συνάδελφο Γιούρι και άλλους για να βρούμε το σωστό ορισμό της καινοτομίας. Και βρήκα εδώ πέρα ένα ορισμό του ΩΣΑ. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους να με ακούσουν, μπορώ να το διαβάσω αν θέλετε, αλλά δεν νομίζω να σας το διαβάσω, θα σας το διανύμω. Ελπίζω όμως ότι θα έχουμε ένα κριτήριο για καινοτομία, για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, ένα κριτήριο το οποίο δεν θα είναι υποχρεωτικό, θα είναι προαιρετικό, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσουμε τις καινοτομίες στην Ευρώπη. Θα στείλω email σε όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους και επειδή το θέμα είναι δύσκολο και περίπλοκο, θα παρακαλούσα, ε, εύχομαι στον Μάκλ και στους σκιώδους συγκητές καλή τύχη. Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Ευχαριστώ. Δεν θα μακρηγορήσω. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για τις ευχές του. Έχουν απομείνει 18-19 ημέρες για να ολοκληρωθεί το θέμα. Ελπίζω όμως να τα καταφέρουμε. Επίσης για την πρόταση περί που έκανε, συμφωνούμε είναι πάντοτε να έχει κανείς έναν ορισμό πάνω στον οποίο να βασιζόμαστε και να μην τα θεωρούμε ως δεδομένα αυτά. Διότι ακόμα και σε ένα δικαστήριο, ε, σε μια δικαστική αρχή μπορεί να υπάρχει προσφυγή και γνωρίζουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα όταν δεν υπάρχουν σαφείς ορισμοί. Δύο γενικές παρατηρήσεις. Υπήρξα μεταξύ εκείνων που ήδη από την αρχή είχα πει ότι αυτό είναι ένας από τους τομεί όπου θα προτιμούσα κατά πολύ να λειτουργούμε με βάση κανονισμό και όχι με βάση οδηγία. Διότι αν υπάρχει μια προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη, στα όσα κάνουμε, θα πρέπει ε, να είναι τα πράγματα ενιαία, απλά, ομοιόμορφα και να έχουν εφαρμογή για όλους. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, συνεπώς ε, πρέπει ε, να δεχθούμε την οδηγία που έχουμε. Αλλά, προφανώς, αυτό το κείμενο δεν θα αλλάξει τον κόσμο. Αντίθετα από το ορισμένοι συνάδελφοι από όλα ε, τα ε, κόμματα έχουν υπενηχθεί. Και το αντιληφθήκαμε όταν προσκρούσαμε ε, στις λεπτομέρειες, στις δυσκολίες των τροπολογιών. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε τον κόσμο εμείς και δεν πρόκειται να απλουστεύσουμε δραματικά τα πράγματα, απλά και μόνο διότι δεν μπορούμε. Επειδή αυτή είναι μια οδηγία και υπάρχουν τόσες ευαισθησίες εθνικής και επαγγελματικής φύσης, είναι προφανές ότι θα επανέλθουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα μοιάζει λίγο πολύ με τα προηγούμενα κείμενα. Ε, θα ήθελα να είναι καλύτερο το δικό μας κείμενο, αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε, αλλά αφού πούμε ειλικρινά ότι δεν πρόκειται να καταφέρουμε ώστε όλα τα δικαστικά συστήματα στην Ευρώπη να είναι τέλεια και πολύ καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα. Δεν θα κατορθώσουμε ε, όλοι οι οργανισμοί προστασίας των ζώων ε, να ε, βελτιωθούν πολύ, ούτε θα λύσουμε το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Ελπίζουμε όμως ότι θα έχουμε επιτύχει κάτι το λογικό. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή υπήρξε πολύ χρήσιμη προκειμένου να ενημερώσουμε το κοινό για το πού βρισκόμαστε και επίσης καταλήξαμε στις συμβαστικές προτάσεις για όλους. Μήπως θέλετε, Κλάσβη, να, μας πείτε ποια είναι η άποψή σας. Στην uh, περιπτώσει χαίρομαι πολύ να ακούσω την άποψή σου σχετικά με το τι πιστεύεις, ποια είναι η άποψή σου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, για την Επιτροπή. Πάντοτε με χαρά βλέπουμε ότι οι προτάσεις μας είναι ένα καλό ξεκίνημα για τις διαπραγματεύσεις και για τον τριμερή διάλογο που ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο. Όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο και η Κορεπέρ πρακτικώς έχουν συμφωνήσει σχετικά με αυτή την οδηγία και ελπίζουμε ότι μπορούμε να πούμε το ίδιο με αυτή την οδηγία για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε γρήγορα με τον τριμερή διάλογο. Για τα συγκεκριμένα θέματα για την απλούστευση, ότι δεν υπάρχει αρκετή απλούστευση. Το πρόβλημα είναι το εξή ότι υπάρχουν πολλά σχετικά με τη μείωση των προδιαγραφών και δημόσιες συμβάσεις, στην διαδικασία διαπραγματεύσεων ή ε, ε, το εργαλείο αυτό. Όλα αυτά δεν καθιστούν πιο ελαφρύ το κείμενο, αλλά επιτρέπουν στις αναθέσεις αρχές να αποφασίσουν αυτό που θέλουν. Γενικά το κείμενο είναι πιο εύληπτο και επίσης είναι σημαντικό επειδή συνιστά κάποια πρόοδο σε σχέση με το υπάρχον κείμενο. Για τη διακυβέρνηση τώρα. Νομίζω ότι ως Επιτροπή είχαμε δεχθεί ότι θα είμαστε υποπτική αρχή, αλλά υπάρχει μια διακυβέρνηση, ένα έργο το οποίο θα πρέπει να παραμείνει για το διαβατήριο των Ευρωπαϊκών Συμβάσεων. Είναι ενδιαφέρουσα πρόταση, αλλά νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει ένα βήμα προόδου και να αναζητήσουμε άμεσα ένα ηλεκτρονικό σύστημα, δηλαδή να μπορεί ένα τέτοιο αρχή να βρει ηλεκτρονικά τα στοιχεία απευθείας από μια βάση δεδομένων, χωρίς να χρειάζεται ο προσφέρον να προσκομίσει κάποιο άλλο έγγραφο ή διαβατήριο, αν θέλετε, οτιδήποτε. Αυτό θα είναι και καλύτερο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις στατιστικές τώρα. Νομίζω ότι αν δείτε το συμβασμό του Συμβουλίου, έχουμε περιοριστεί στο ελάχιστο και πρέπει να καταλάβουμε όμως πώς λειτουργεί η αγορά. Τέλος, κατελήγοντας, θα ήθελα να πω δύο-τρία λόγια για θέματα που δεν συζητήθηκαν σήμερα. Προφανώς προσπαθούμε να, ακολουθεί, να δούμε τις συμβαστικές τροπολογίες, αλλά μας απασχολούν ορισμένες τροπολογίες και συμβασμοί, επειδή έχουμε την εντύπωση ότι ακόμα και εδώ δεν, δεν είμαστε όσο φιλική προσωπική αγορά, δεν είστε τόσο φιλική προσωπική αγορά όσο το Συμβούλιο ε, και η Επιτροπή. Πιστεύουμε ότι η διαφάνεια είναι κάτι το απαραίτητο αν θέλουμε να λειτουργήσει το σύστημα. Το δεύτερο θέμα είναι το θέμα της ε, συνεργασίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπου πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι σαφής ε, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ, συνεργασία μεταξύ δημοσίων αρχών και ότι αυτό πρέπει να αναφερθεί στο κείμενο. Διαφορετικά θα υπάρχει νομική ασάφεια και δεδομένου ότι αυτή η συνεργασία στο δημόσιο τομέα είναι σημαντική, πρέπει να είναι απόλυτα σαφής. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Ταραμπέλα, σύντομα μια ανακεφαλαίωση, γιατί αύριο το πρωί θα ξαναλάβετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φυσικά θα είμαι σύντομο, επειδή έρχεται η ώρα τη ψηφοφορία. Ακούγοντα όμω όλα αυτά τα σχόλια, θα προσπαθήσω να συνοψίσω, αλλά κάτι το οποίο επαναλήφθηκε συχνά είναι ότι λυπούνται οι παρεμβαίνοντε που δεν υπάρχουν μεγαλύτερε απλουστεύσει. Αυτό το οποίο είπατε εσεί, κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό όταν είπατε ότι η απλούστευση, το κλειδί για την απλούστευση είναι η ασφάλεια των κανονισμών, των κανόνων. Και όταν προσθέτουμε έννοιες δεν σημαίνει ότι τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκο, αλλά θέλουμε να έχουμε ένα κανόνα σαφή, ένα, μια εργαλειοθήκη, ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε ή όχι, ο καθένας κατά βούληση θα αποφασίσει και όπως είχε πει ο κ. Σουάπ με πολύ σκεπτικισμό, αλλά μπορούμε να είμαστε σκεπτικοί. Το θέμα είναι να μην είμαστε ευρωσκεπτικιστές και να φροντίσουμε ώστε πέραν από τις έννοιες που υπάρχουν και η Επιτροπή άρχισε να αναφέρει νέε έννοιε στην πρόταση τη του Δεκεμβρίου 2011, προσθέτει νέε έννοιε. Αλλά φυσικά δεν είναι τόσο εύκολη η απλούστευση. Αυτό που θα έλεγα όμω είναι μπορούν, τα πράγματα είναι πιο απλά. Αρκεί να πούμε ότι η χαμηλότερη τιμή γενικεύεται, ε, δεν λαμβάνει υπόψη τα περιβαλλοντικά κριτήρια, τα κοινωνικά κριτήρια. Έχουμε μία διαδικασία, η οποία είναι μια διαδικασία που δεν δημοσιοποιείται, ε, γίνεται τη διαπραγμάτευση, αλλά δεν υπάρχει δημοσιοποίηση. Τα πράγματα είναι πιο απλά, αλλά δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια, λιγότερο ανταγωνισμό, δεν υπάρχει επιλογή για τι δημόσιε αρχέ να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν την πιο ε, συμφέρουσα οικονομική προσφορά. Αλλά όπω είπε και ο Επίτροπο ο κ. Μπαρνιέ, είπε ότι μέσα από αυτή την οδηγία τι πρέπει να γίνει το 19% του ΑΕΠ που αντιπροσωπεύει δημόσια παραγγελία στην Ευρώπη να επενδύεται με πιο αποτελεσματικό τρόπο ε, εξυπηρετώντας την Ευρώπη και τους πολίτες ε, με γνώμονα την βιωσιμότητα. Είναι γεγονός και στη Γεωργία σημαίνει αυτό. Εγώ τώρα ασχολούμαι με την κοινή αγροτική πολιτική υπάρχει μια έκθεση πρωτοβουλία ε, και εκεί μέσα μπορεί κανεί να αναφέρει γενικέ αρχέ που μα βρίσκει όλου σύμφωνου και η έκθεση κυρία Ρούδαν το αποδεικνύει θαυμάσια έκθεση με πολλέ νέε έννοιε. Όλα πολύ καλά. Όταν όμω θέλουμε να μεταφράσουμε τι έννοιε σε νομοθετική πρόταση, τα πράγματα περιπλέκονται. Το ίδιο συμβαίνει με την ΚΑΠ. Είχαμε μια θαυμάσια έκθεση του κ. George Λάιεν, του κ. Λεφόλ, του κ. Μποβέ. Θαυμάσιε εκθέσει την ε, ε, γραπτή έκθεση του κ. Ντες και όταν φτάνει κανείς ε, στις αποφάσεις για την κοινή ερωτική πολιτική, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα και καμιά φορά έχουμε την τάση να μην τηρούμε τις αρχές μας. Τώρα, Ω προ τι τροπολογίε, δεν μπορώ τώρα να δώσω απαντήσει, επειδή η κυρία Ρούλα έκανε πολλέ σκέψει για το διαβατήριο αυτό. Ήθελα να πω ότι αυτό το διαβατήριο είναι και ένα πλεονέκτημα. Το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο είναι το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται κανείς να προσκομίζει εκ προημίου πολλά έγγραφα. Ε, οι επιχειρήσει έπρεπε να προσκομίζουν πολλά πολλά έγγραφα που ήταν, που ήταν άχρηστα. Σήμερα το διαβατήριο επιτρέπει ε, με μια επιστοποίηση να ε, συμμετέχει κανείς σε διαγωνισμούς, σε δημοπρασίες και εκείνο στο οποίο κατακυρώνεται το έργο να προσκομίσει τα συμπληρωματικά έγγραφα που του ζητούνται. Το διαβατήριο λοιπόν ήταν μια μορφή απλούστευση. Τώρα, Άλλε έννοιε. Ο κ. Δεγιόν μίλησε για το άρθρο 15. Απλά θέλω να σας πω ότι στην αγγλική εκδοχή υπάρχει αυτή η λέξη το where applicable ε, ενώ είχε συμφωνηθεί θα διαγραφεί το where applicable όπου ισχύει. Νομίζω ότι αυτό λησμονήθηκε. Για τον κύριο Παλασάρε, ναι. Βραμέτα Πεκάρο. Είναι κρίμα, αγαπητοί συνάδελφοι, που δεν θα παραστείτε αύριο στη συνεδρίαση. Μακάρι να μπορούσα να αναβάλω και εγώ την πτήση σας, αλλά δεν γίνεται. Κύριε Βαντέρς, αγαπητέ συνάδελφε, η καινοτομία, συνεχίζω γαλλικά, γαλλικά, η καινοτομία. Ειλικρινά, θαυμάσια είναι αυτά που λες, αλλά είσαι εισηγητής στην Επιτροπή και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή η Επιτροπή ε, σκιώδης εισηγητής ότι υπογραμμίζει αυτή η Επιτροπή την ε, σημασία να υπάρχουν κριτήρια, όχι μόνο περιβαλλοντικά δουλειά σα είναι, αλλά και κοινωνικά κριτήρια. Νομίζω ότι ίσω ξέχασε να το αναφέρει, αλλά η έκθεση της Επιτροπής μας ε, εντυπωσιάστηκα πολύ από αυτή την ε, έκθεση τη Επιτροπής και από άλλε. Ο Φρονκ Άγγελ έλεγε να μην αλλάξουν όλα. Και θα έλεγα ευτυχώ που δεν αλλάζουμε όλα. Γιατί Υπάρχουν πράγματα που πάνε καλά στι δημόσιε συμβάσει. Ε, υπήρχαν οι δύο οδηγίε το 17-18-2004 όπου οι χώρε ε, φύρμωσαν με δυσκολία τα κεκτημένα αυτών των ιδιών αλλά ένα μεγάλο μέρο των δημοσίων αγορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο λειτουργεί πολύ καλά. Και καταλήγω πρόεδρε λέγοντα ότι ίσω, ε, δεν με χειροκροτήσατε, μπορεί στις 18 Δεκεμβρίου να με χειροκροτήσετε, ή τον Ιανουάριο. Εν πάση περιπτώσει όμως ε, κάτι ήταν μια σταθερά και το ότι χαιρετήσατε το έργο όλων όσων συνέβαλαν σε αυτή την έκθεση, στους οικειώδεις συγητές, τους οποίους ευχαριστώ λόγω της δουλειάς που έκαναν, ε, την γραμματεία της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ, ε, το προσωπικό των πολιτικών ομάδων και επιτρέψατε μου ότι και εγώ δούλεψα με την Σαρτίνα Πλάι εδώ από την σοσιαλιστική ομάδα και την Αλέτσια ε, Τσενκιόνη, τη βοηθό μου, χωρίς αυτά τα, αποτελεσματικά άτομα, τα δραστήρια άτομα, δεν θα ήμασταν τίποτα εμείς και δεν θα είχαμε ένα έγγραφο το οποίο ελπίζω θα βελτιώσει ε, την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Good. Well, thank you very much. It's been a very good... Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση. Και όπως είπατε και εσείς, Αύριο θα κάνουμε συνάντηση και κλεισμένο των θυρών για τις διαπραγματεύσεις, αλλά προφανώς ε, είναι προσκεκλημένα όλα τα μέλη της Επιτροπής, αν το επιθυμούν. Δεν είναι και κλεισμένο των θυρών για τα μέλη της Επιτροπής. Λοιπόν, όσοι αποχωρούν, ας αποχωρήσουν ησύχως παρακαλώ. Και αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, όπως είπε και ο κ. Σταραμπέλα Κύριε Μάντερς, παρακαλώ, κύριε Μάντερς. Τώρα πρέπει να πάμε στην ψηφοφορία. Ήσυχα αποχωρήστε παρακαλώ. Να σκεφτούμε λίγο αυτό που είπε ο κύριος Ταραμπέλα, ότι δεν είναι απλή υπόθεση η απλοποίηση. Αλήθεια είναι αυτό. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε το χρόνο των τριών εβδομάδων. Λοιπόν, τώρα θα ψηφίσουμε. Ενεργειακός χάρτης πορείας είναι το πρώτο για το 2050. Είναι η έκθεση του κυρίου Σμιτ, ο οποίος επίσης δεν είναι παρόν. Δεν ξέρω ποιος από την ομάδα των φιλελευθέρων θα κάνει την παρουσίαση. Ποιος θα το παρακολουθήσει. Θέλετε κάποιους. Α, προχωράμε κατευθείαν. Δεν χρειάζεται. Όλες οι συμβαστικές είναι ξεκαθαρισμένες. Πάμε στην ψηφοφορία κατευθείαν. Είμαστε λοιπόν στην έκθεση ΣΜΙΤ, Ενεργειακός Χάρτης Πορείας για το 2050, γνωμοδότηση, ε, ε, 1 υπέρ. Ας ε, ελέγξουμε το σύστημα, να δούμε και ποιος είναι εδώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 1. «35 είναι, όχι 36. Υπάρχει άλλος που έχει ε, κάρτα. Πέρας τη ψηφοφορία. Μάλιστα. 18 προς 18. Ε, δεν ε, γίνεται δεκτή. Πάμε στην τροπολογία 2. Α, πολύ αργά. Δεν με ακούσατε έγκαιρα. Επόμενο, ψηφίζουμε την τροπολογία 2 υπέρ. Κατά δεκτή. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Πάμε τώρα στην τροπολογία 7 του κυρίου Χέντλε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, στην τροπολογία 7. Υ, ε, υπέρ. Κατά. Απερίφθη. Κυρία Βέσνα. Είστε υπεύθυνοι... Α, δίνετε το... για τη ομάδα σοσιαλιστών... Μάλιστα. Για να ξέρω αν θα γίνει ψηφοφορία. Τροπολογία 8. Ε, υπέρ. Κατά. Σαφώς δεκτή. Τροπολογία 9. Καταπίπτει νομίζω. Α, ως προσθήκη. Ε, τροπολογία 9 ως προσθήκη. Υπέρ υπέρ, κατά, σαφώς υπέρ, συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, δεκτή, 27 υπέρ, κατά, δεκτή, η τροπολογία 10 υπέρ, κατά, δεκτή, η 11 υπέρ, κατά, δεκτή, 14 υπέρ, κατά δεκτή, 15 υπέρ κατά δεκτή, 16 υπέρ κατά σαφώς δεκτή, η 18 έχει αποσυρθεί. Πάμε στη συμβιβαστική 4 υπέρ κατά σαφώς δεκτή, συμβιβαστική 5 υπέρ κατά δεκτή. Πάμε τώρα στην 26. Έτσι δεν είναι, μάλιστα. 26 υπέρ, κατά, ε, δεκτή. 29. 29. Έχουμε εδώ, δίνεται, α, ελεύθερη, ε, κατά συνείδηση ψήφος. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Θα καταγράψουμε την ψήφο κατά τη δική σας. Ψηφίζουμε την 29. Κάποιος δεν ψήφισε, αλλά εγώ είπα πέρας. Μάλιστα. 22 είναι κατά. κατά. Έχει απορριφθεί. Τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Δεκτή σαφώ. 31. Υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 33. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 34. Τμηματική ψηφοφορία. χωρίς τη λέξη εθνικός, υπέρ, κατά, δεκτή. Και το δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Πέρας. 19 υπέρ, 18 κατά, δεκτή. Η τροπολογία 35 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 36 αποσύρθηκε 6 υπέρ συμβαστική κατά αποχές δεκτή τροπολογία 39 του κυρίου Ιέ της κυρίας Μπάστος υπέρ κατά δεκτή 44 επίσης της κυρίας Μπάστος κατά δεκτή τροπολογία 40 υπέρ κατά δεκτή 45, τμήματική ψηφοφορία. Βλέπετε το πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά, δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Πέρας. Δεκτό. 19 υπέρ 17 κατά. Και μια αποχή. 48 υπέρ. Κατά δεκτή. 43 έχει καταπέσει λόγω της συμβιβαστική. Πάμε στην 46. Υπέρ. Κατά δεκτή σαφώς. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία επί των τροπολογιών και άρχεται η ψηφοφορία επί του... της γνωμοδοτήσεως. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Ναι, έχω 34. Μήπως δεν ψήφισε, δεν κανείς. Έχουν κάποιοι κάρτες και δεν... Όχι, τώρα, τώρα ψήφισαν όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 32 υπέρ. 4 κατά χωρίς αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Σμιτ εν τη απουσία του. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα προχωρούμε σε μια δεύτερη γνωμοδότηση βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση που είναι του εισηγητού μας του κυρίου Χατζημαρκάκης, λείπει και εκείνος. Θέλει κανείς να μιλήσει εξ ονόματός του, ναι, όχι, όχι. Ο, καλώς, πάμε στην ψηφοφορία κατευθείαν. Τροπολογία 1 της κυρίας Χάντσλικ, υπέρ. Κατά, αποχές δεκτή, συμβιβαστική 1 υπέρ κατά δεκτή, συμβιβαστική 2 υπέρ κατά δεκτή, 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 6 ως προσθήκη υπέρ κατά δεκτή, σε 7 ως προσθήκη υπέρ κατά απερίφθη αυτή. Τροπολογία 8 υπέρ. Υπέρ παρακαλώ να δω καλά. Κατά. Σαφώς δεκτή. Τροπολογία 9. Όχι, αυτέ 9 και 10 καταπίπτουν. Πάμε στην 11 του κυρίου Ούμπερμαϊρ. Εδώ πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά νομίζω. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 11. Πέρας. 22 υπέρ 15 κατά. Τροπολογία 12 υπέρ κατά δεκτή. Τροπολογία 13 υπέρ κατά δεκτή και αυτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά δεκτή. 15 της κυρίας Μακλάρκιν υπέρ κατά δεκτή. 16 υπέρ κατά Δεκτή 17 υπέρ κατά δεκτή και αυτή. Η 18 προσθήκη υπέρ κατά δεκτή. 19 υπέρ κατά δεκτή. 20 του κυρίου Ομπερμαϊρ υπέρ κατά απερίφθη. 21 υπέρ κατά δεκτή 22 υπέρ κατά δεκτή 23 υπέρ κατά δεκτή 24 υπέρ κατά δεκτή 25 25 υπέρ κατά δεκτή 26 υπέρ κατά δεκτή και αυτή. 27 υπέρ κατά δεκτή συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή 33 υπέρ κατά νομίζω ότι θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά εδώ στην 33 ψηφίζουμε την τροπολογία 33 άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή 20 προς 16 και 34 υπέρ κατά δεκτή σαφώς και τώρα άρχεται η ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου γνωμοδοτήσεως. Άρχεται η ψηφοφορία. Κατεβήκαμε στους 35. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή. 34 υπέρ. 35 ψήφοι υπέρ. Μία ψήφος κατά. Σημειώσαμε την κυρία Κανέτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν για την ε, καλή διεξαγωγή της ψηφοφορία. Ευχαριστούμε. Right. So we'll just let everyone leave. Βλέπω ότι φεύγουν όλοι, μην φύγετε όμως.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 Uh, I'm just allowing a bit of a short break because I think. Uh, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Γιατί περιμένουμε νομίζω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κάνει μια παρουσίαση. Να περιμένουμε κυρία Κοράτσα Μπίλτε. Okay. Do you want to... Um, uh, Anna Maria, do you want to introduce Αναμαρία, μήπως θέλετε να κάνετε μια σύντομη εισαγωγή. Um, Ωραία λοιπόν. Είναι ακριβώς 4 και μισή. Δεν θα ήθελα να καθυστερήσουμε άλλο, γιατί μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που θα μπαίνουν στο διαδίκτυο για να παρακολουθήσουν την παρουσίαση της Άννας Μαρίας για τις ε, ε, υπηρεσίες της εσωτερικής αγοράς ε, ε, την εσωτερική αγορά υπηρεσιών, να καλωσορίσω και μια ομάδα ε, επισκεπτών από την Σουηδική Ένωση Επιχειρηματιών. Ήρθαν ενώ έλειπα, καλωσορίσατε λοιπόν και ελπίζω να συμμετέχετε και εσείς στη συζήτηση, ε, να σας ενδιαφέρει δηλαδή το ζήτημα για το όλο ζήτημα της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών Είχα συναντήσει μέλη της Επιτροπής σας το 2009 στη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας και υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε μια έκθεση δύο πρωτοβουλίας για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών, την περιγραφή της κατάστασης και τα επόμενα βήματα Ελπίζω η Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς κάνουν αυτοί, ιδίω σε σημαντικούς τομείς, όπως για παράδειγμα την αμοιβαία αξιολόγηση των περιορισμών μεταξύ των κρατών μελών, ε, για σημεία επαφής και αντίστοιχα ζητήματα. Αλλά καταρχάς να δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλτ, για να μας παρουσιάσει λίγο ε, το σκηνικό, αν θέλετε, και μετά θα ακούσουμε την κυρία Φρασφάνς Πανσέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άννα Μαρία λοιπόν να μας πει λίγα εισαγωγικά πράγματα και από εκεί και πέρα θα επανέλθουμε στη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε σας ευχαριστώ που καλωσορίσατε και τους επισκέπτες μας. Φαίνεται να έχουμε εδώ τους ανθρώπους που πραγματικά δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά και γι' αυτό πρέπει να τους δώσουμε και απαντήσεις. Γιατί δύο χρόνια μετά από την προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας για τις υπηρεσίες που έγινε το 2009, εγκρίθηκε το 2006, εξακολουθούμε να έχουμε την πλειονότητα των κρατών μελών χωρίς να έχουν εφαρμόσει πλήρως ή να έχουν μεταφέρει σωστά την οδηγία για τις υπηρεσίες. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητήθηκαν πληροφορίες σε 26 κράτη-μέλη, 27 είμαστε όλοι και όλοι. Και απέστειλαν 26 επιστολές ε, για πληροφορίες και από αυτές τις επιστολές οι 21 επιστολέ ήταν για την οδηγία για τις υπηρεσίες και στις 21 αυτές οι επιστολές έλαβαν θετικές απαντήσεις μόνο σε τέσσερις. Καλό μεν, αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 16 κράτη-μέλη με σαφείς διαδικασίες επί παραβάση και πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως οι διαδικασίες. Αυτό καταδεικνύει γιατί είναι τόσο σημαντική η εξέταση αυτής της ε, οδηγίες για τις υπηρεσίε, και γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι τιμή μου που μου αμαθέσατε αυτή την έκθεση στο Κοινοβούλιο. Έχουμε μια πολύ καλή βάση ως κίνηση, διότι έχουμε ε, δύο εξαιρετικέ εκθέσεις για την εφαρμογή τη οδηγία για τις υπηρεσίε και για την αμοιβαία αξιολόγηση τη οδηγία για τις υπηρεσίε. Αυτό σημαίνει ότι ε, θέσαμε τους στόχους και καθορίσαμε ε, πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε και τώρα χρειαζόμαστε απλώς την πολιτική όθεση ώστε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν χρησιμοποιούνται κάθε μέρα ε, τα όσα μας προσφέρει η οδηγία για τις υπηρεσίες. Θέσεις εργασίας, ωφέλη για τους καταναλωτές. Και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας, και με τους κοιόδης συζητητές και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά και τους ενδιαφερομένους, προκειμένου να μπορέσουμε να διαβιβάσουμε ακριβώς αυτό το μήνυμα. Κάποιοι θεωρούν ότι το να υπερβούμε την κρίση γίνεται μόνο εάν κλείσουμε τις, τους ορίζοντές μας. Και πραγματικά ε, πιστεύω ε, ότι θα πρέπει να με υποστηρίξετε για να πείσουμε τον κόσμο ότι για να ξεφύγουμε από την κρίση πρέπει να ανοίξουμε τις υπηρεσίες μας. Οι υπηρεσίες είναι το 65% των θέσεων εργασία Είναι το 70% της συνολικής απασχόλησης στην Ευρώπη, μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ μας, το 6,5% και η πλήρης λειτουργία της εσωτερικής αγοράς δεν υπάρχει εάν δεν εφαρμοστεί όπως πρέπει η οδηγία για τις υπηρεσίες. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι το βασικό πολιτικό μήνυμα που θα πρέπει να αποστείλουμε στα κράτη-μέλη, ιδίω σε περίοδο κρίση. Επιτέλους λοιπόν κατανοήσαμε και βρίσκεται πλέον και στο επίκεντρο της συζήτησης το γεγονός ότι δεν μπορούμε να δαπανούμε συνεχώς, δεν έχουμε δημόσια κονδύλια και επομένως πρέπει να δημιουργήσουμε ανάπτυξη, θέσεις εργασία και να συνεχίσουμε να είμαστε και πιο ανταγωνιστικοί απελευθερώνοντα το δυναμικό της ε, ε, ενίας αγοράς. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι πραγματικά δυνατότητα ανάπτυξης, είναι οι υπηρεσίες στην Ευρώπη. Έχουμε μια εξαιρετική βάση εργασίας λοιπόν η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσβλέπω και στα περισσότερα που έχετε να μας πείτε, αλλά θα ήθελα ε, να πω ότι οι βασικές γραμμές με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνοι. Μηδενική ανοσυχή στις παρατυπίες για την οδηγία για τις υπηρεσίες. Και επίσης θα ήθελα εδώ να αποτίσω φορό τιμής και στον Επίτροπο Μπαρνιέη, διότι έκανε τον κόπο να πάει σε κάθε κράτος μέλος και να μιλήσει πραγματικά με τους ενδιαφερομένους για την εφαρμογή της οδηγίας για την της να δει ποια είναι τα ε, θέματα που τους απασχολούν, τα σημεία επαφής και προσπάθησε ε, να μεταφέρει εδώ στις Βρυξέλλες τα όσα έμαθε από τα 27 κράτη-μέλη. Να σας πω σε τι αναφερόμαστε. Αρχιτέκτονες, παραδείγματι, που για να ε, ξεκινήσουν μια επιχείρηση σε ένα κράτος μέλος χρειάζονται ένα αρχικό κεφάλαιο, και πρέπει κατά 51% να επανδρώνονται από ε, ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό ουσιαστικά επιβάλλει ένα επιχειρηματικό μοντέλο σε ένα τεράστιο επαγγελματικό κλάδο. Ε, υπάρχουν κάποιες ε, δυνατότητες ε, προστιθέμενης αξίας για να δραστηριοποιηθεί κάποιος σε ένα κράτος μέλος. Υπάρχουν, για παράδειγμα, νομικές απαιτήσει, επιπλέον αδειοδοτήσει για να ξεκινήσει κάποιος να εργάζεται σε άλλη χώρα. Αλλά ένα στοιχείο που προκύπτει και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε είναι ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες αιτήσει από τους καταναλωτές καταναλωτές που δεν μπορούν καν να ε, κατεβάσουν το Spotify ή το iTunes ε, ε, εντός της εσωτερικής αγοράς. Υπάρχουν αναφορές από καταναλωτές διότι αν αγοράσει κάποιος ένα πακέτο για μια κρουαζιέρα σε ένα κράτος μέλος πληρώνει μία τιμή και αν είσαι πολίτης άλλης χώρας πληρώνει το διπλάσιο. 1.200 ευρώ ο ένας, 2.400 ο άλλος. Ε, και πραγματικά θα ήθελα να ζητήσω από όλους να διαβάσει το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δίνει πάμπολα τέτοια παραδείγματα. Διότι πρέπει να περάσουμε πλέον στη δράση για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία διαπιστώνουμε. Κύριε Πρόεδρε, περιμένω να ακούσω και πολλά περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι σκοπεύει να κάνει από εδώ και στο εξή. Νομίζω ότι η άποψή τους ε, να έχουν μια δεύτερη γενεά ε, σημείων επαφής είναι πολύ σημαντικό διότι η οδηγία για τις υπηρεσίες ε, και ο κόσμος των υπηρεσιών γίνεται όλο ένα και πιο ψηφιακός, επομένως χρειαζόμαστε και ψηφιακές πλατφόρμες για να δίνουμε πληροφορίες ε, σε όσους δραστηριοποιούνται μέσω υπηρεσιών στην ενιαία αγορά. Θα σταματήσω τώρα λοιπόν για να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους και να ακούσω τις απόψεις τους και θα ήθελα στη συνέχεια κύριε Πρόεδρε να μου δώσετε το λόγο για να ολοκληρώσω τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ σαφή παρουσίαση. Η ιδέα είναι ότι μπορούμε να ζητήσουμε κ. να εξηγήσει τι κάνει η Επιτροπή. Έχαμε ανακοίνωση και τα κείμενα και κατόπιν θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα μεταξύ μας θα είναι ένα καλό πλαίσιο. Και επίσης υπάρχει και μία ακρόαση. Αυτά όλα μπορούν να συζητηθούν σε σχέση με το τι πρέπει να κάνουμε. Ε, χαιρετίζω λοιπόν, καλωσορίζω την ομάδα της ε, Επιτροπής, και, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, σχετικά με το έργο του κ. Μπαρνιέ. Και τους ευχαριστώ, σημειώνω όμως, ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή οι Πρωθυπουργοί και Αρχηγοί Κρατών υποστηρίζουν αυτή την έκθεση που δείχνει ότι υπάρχει πολιτική στήριξη. Και γι' αυτό... Thank you, Mr. Chairman. Um, so on the... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις 8 Ιουνίου η Επιτροπή υιοθέτησε μία ανακοίνωση για μια εταιρική σχέση, για νέα ανάπτυξη των υπηρεσιών, ε, συνοδευόμενα με τρία έγγραφα του προσωπικού. Η μία που υποστήριζε την οδηγία τη υπηρεσία Δεύτερον, αυτό το οποίο ονομάζουμε του ελέγχου αποδόσεων για τους τρεις βασικούς τομείς ε, της οικονομίας, οικοδομή, τουρισμό και οι επιχειρητικέ υπηρεσίες και πώ υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των νέων νομοθεσιών και η καθοδήγηση τη οδηγία που απαγορεύει ε, την διάκριση ε, αποδεκτών υπηρεσιών με βάση την υπηκότητα και την, τον τόπο διαμονής. Θα υπογραμμίσω τώρα ποια είναι τα σχέδιά μας σε σχέση με το καθένα. Όσον αφορά την οδηγία των υπηρεσιών, υπάρχουν τέσσερα μεγάλα κεφάλαια. Το πρώτο, όπως ανέφερε η προλαΐσασα, μηδενική, η πολιτική τη μηδενικής ανοχής. Θα έπρεπε να πω αρχικά ότι η οδηγία των υπηρεσιών μεταφέρθηκε και στα 27 κράτη-μέλη και οδήγησε σε περισσότερα από χίλια νομοθετήματα. τροποποιήθηκε, αναθεωρήθηκε, ανασυντάχθηκε, υιοθετήθηκε τελικά και σε γενικές γραμμές εφαρμόστηκε αρκετά καλά. Πέρσι μελετήσαμε την εφαρμογή και υπάρχουν υποχρεώσεις που πηγάζουν από την οδηγία, όταν υπάρχει διακριτική ευχαίρεια από τα κράτη-μέλη. Σε αυτές τις ε, περιπτώσεις ε, η εφαρμογή δεν ήταν πολύ καλή. Γι' αυτό αυτά τα θέματα ε, τα θίγουμε σε επιστολές μηδενικής ανοχής που στείλαμε στα κράτη-μέλη και υπάρχουν ορισμένε διαδικασίες πριν από τις παραβάσεις σε 12 περιπτώσεις. Αυτή ήταν η, το πρώτο σκέλος της εργασίας μας. Το δεύτερο είναι να οθήσουμε τα κράτη-μέλη να ξεπεράσουν την αμυγός νομική εφαρμογή ε, της οδηγίας και να λάβουν υπόψη τις οικονομικές επιπτώσεις της οδηγίας. Κυρίως λαμβάνοντας υπόψη δύο στοιχεία. Το πρώτο, τις απαιτήσεις, ε, ε τις νομικές απαιτήσεις και τις πάγιες τιμές που ορισμένα Σταθερέ τιμέ που θα πρέπει να εφαρμόσουν ορισμένοι επαγγελματίε. Επίσης, η ελευθερία παροχής υπηρεσιών, που είναι βασικά η δυνατότητα να παράσχει κανεί υπηρεσίες διασυνοριακά ε, και σε προσωρινή βάση, σε αντιδιαστολή με την εγκατάσταση σε ένα κράτος μέλος. Αυτό θα το κάνουμε χρησιμοποιώντα κυρίω την αθεώρηση των νομοτήμων από τα κράτη-μέλη, που θα ξεκινήσει στα μέσα Δεκεμβρίου και θα επεκταθεί μέχρι την Άνοιξη. Η ιδέα είναι ότι θα πρέπει να σωματωθεί ε, στο Ευρωπαϊκό ε, Εξάμεινο του 2013 και αν παραστεί ανάγκη, ανάλογα με τα αποτελέσματα της ε, αναθεώρησης από τους ομοτήμους, μπορεί να καταλήξουμε σε νέα νομοθεσία. Αυτή η αναθεώρηση από τους ομοτήμους θα εστιαστεί σε επιλεγμένες δραστηριότητες και δεν μπορούμε να έχουμε πολύ ευρύτατο πεδίο, πολύ ευρύ πεδίο εφαρμογής. Αυτή η αναθεώρηση από σωματήμους συνίσταται σε ομάδες 8 ή 9 ε, ατόμων στα κράτη-μέλη και αυτές οι ομάδες θα παραβάλλουν τα συστήματά τους. Το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να είναι σαφές και θα γίνει με βάση πέντε επιλεγμένες δραστηριότητες περιλαμβανομένων και των αρχιτεκτών αλλά και τους λογιστές, ε, τους κτηνιάτρους κλπ. Όσον αφορά την, την ρήτρα της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες ανάμεσα στον πάροχο της υπηρεσίας που θέλει να εγκατασταθεί και σε εκείνον ο οποίος επιθυμεί μόνο να παράσχει υπηρεσία σε προσωρινή βάση. Αυτή η διαφορά δεν είναι πάντοτε σαφής, το οποίο σημαίνει ότι ο πάροχος υπηρεσίας, ο οποίος νομικά είναι εγκατεστημένο σε μια χώρα, μπορεί να κληθεί να πληρεί πολύ αυστηρέ προποθέσει όταν θα μεταβεί σε ένα κράτο μέλο μόνο για να παράσχει προσωρινώ υπηρεσίε. Ενώ στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε να υπόκειται σε απαιτήσει ή σε όρου ή τουλάχιστον σε ελάχιστε απαιτήσει σε σχέση με εκείνου που έχουν εγκατασταθεί σε εκείνη τη χώρα. Αυτό είναι ένα θέμα αμφιλεγόμενο και θα το δούμε με τα κράτη-μέλη ως προς τη μεγιστοποίηση των οικονομικών επιπτώσεων της οδηγίας ε, υπηρεσιών. Αυτό είναι το, το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι τα θέματα ασφάλειας. Ε, όσον αφορά την διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, οι παροχή υπηρεσιών ουσιαστικά θέλουν να παρέχουν υπηρεσίες σε προσωρινή βάση σε άλλο κράτος μέλος και εκεί αντιμετωπίζουν δυσκολίες να βρουν έναν ασφαλιστή ή πρέπει να πληρώνουν πολύ ψηλά ασφάλιστρα για να ασφαλιστούν. Και αυτό συχνά είναι ένα κόλλημα. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δούμε τι θα γίνει με τον ασφαλιστικό κλάδο και να καταλήξουμε σε μια έκθεση το 2013 με τις δυσκολίες που θα παρουσιάσουμε και τελικά θα προτιμούσαμε να βρούμε λύσεις με βάση τους διάφορους τομεί, δηλαδή πρακτικές λύσεις ανάλογα με τι περιπτώσεις. Υπάρχουν πολλοί όμιλοι ε, ασφαλιστικών εταιριών, υπάρχουν εταιρικέ σχέσεις, συμπράξει μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών ε, στα διάφορα κράτη-μέλη και η βασική ιδέα είναι να προωθήσουμε, να προαγάγουμε ρεαλιστικέ λύσει. και στις δύο περιπτώσεις θέλουμε μηδενική ενοχή να μεγιστοποιήσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις και οικονομικά ωφέλη πέρα από το γράμμα ε, ε της οδηγίας των υπηρεσιών. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα ωφελήσει τους καταναλωτές αυτή η οδηγία. Και το άρθρο 20 παράγραφος 2 που απαγορεύει τη διάκριση ε, των αποδεκτών ε, των υπηρεσιών με βάση τη διαμονή ή την υπηκότητα. Εκείνο το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να δούμε μαζί με τους εθνικούς θεσμούς που είναι υπεύθυνοι, αρμόδιοι για την εφαρμογή αυτού του άρθρου, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς εφαρμόζουν αυτούς τους κανόνες και η ιδέα είναι μέχρι το τέλος του 2013 να τους δώσουμε περισσότερες οδηγίες σχετικά με το πόσο ε, θα εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα και το 2013 θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση μεταξύ των καταναλωτών, διότι πρέπει οι καταναλωτές να καταλάβουν αν η Ευρώπη υπάρχει ή δεν υπάρχει. Για αυτούς είναι πολύ σημαντικό και συνεπώς αυτή η δεν υπαρχει Γι' αυτους είναι ιδιαίτερα σημαντική το, η τελευταία μας γραμμή είναι αυτά τα σημεία επαφής, το ενιαίο σημείο επαφής. Δηλαδή, η πάροχη υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σε θέση μέσω ενός ενιαίου σημείου επαφής να βρουν όλες τις πληροφορίες που έχουν σχέση με την οδηγία των υπηρεσιών και την παροχή υπηρεσιών σε μια άλλη χώρα και ενδεχομένως να είναι σε θέση να εφαρμόσουν όλες τις διαδικασίες διαδικτυακά. Τα κράτη-μέλη κατέβαλαν προσπάθειες. Οι προσπάθειες όμως δεν έχουν αποδώσει παντού. Ε, δημοσιεύσαμε μια μελέτη σχετικά που καταδεικνύει ότι ορισμένες χώρες έχουν προχωρήσει πολύ, άλλες ε, είναι καθυστερημένες σε αυτό το δομέα και άλλες κάπου στη μέση. Προσπαθήσουμε να τους προωθήσουμε με βάση τρία στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, να θέλουμε το σημείο ενιαία επαφή να ξεπεράσει αυτή την οδηγία υπηρεσιών και να καλύψει όλο τον επιχειρησιακό κύκλο. Αυτό το εργαλείο για να είναι χρήσιμο σε έναν πάροχο υπηρεσιών θα πρέπει να ε, περιέχει όλες τις πληροφορίες ε, που τον ενδιαφέρουν και όχι μόνο πληροφορίε που βρίσκει ήδη στην οδηγία υπηρεσιών, οι οποίε κατά την άποψή του είναι πολύ γενικέ. Το δεύτερο, αυτό το ενιαίο σημείο επαφή πρέπει να είναι πολύγλωσσο τουλάχιστον δίγλωσσο, σε μία γλώσσα που είναι κατανοητή από του περισσότερου πολίτε. Και το τελευταίο σημείο θέλουμε να είναι πιο φιλικό προς το χρήστη, δηλαδή ε, για έναν πάροχο υπηρεσιών να είναι ευνόητο, να μπορεί να βρει τι πληροφορίε που θέλει εύκολα. Και κατόπιν ε, να είναι ρεαλιστική προσέγγιση, ε, θα δοκιμάσουμε αυτά τα ενιαία σημεία επαφής η μελέτη η οποία διενεργήθηκε για τις οικονομικές επιπτώσεις στις οδηγίες υπηρεσιών μας δείχνει ότι το 0,27% του ΑΕΠ μπορεί να κερδιθεί εάν λειτουργήσουν καλά αυτά τα νέα σημεία επαφής. Είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Και κατόπιν ε, ένα διετές σχέδιο για να παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε αυτό το τομέα. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία. Υπάρχουν και άλλα θέματα, τα οποία δεν θα σας αναφέρω τώρα, εκτός αν θέλετε να επισέλθω σε λεπτομέρειες, θέματα που αφορούν ε, τα επαγγελματικά προσόντα και την σχετική οδηγία που αφορά τις ανάγκες ορισμένων συγκεκριμένων τομέων, όπως ε, λιανικός τομέας, εξειδικευμένες υπηρεσίες, αλλά φαντάζομαι ότι η κυρία η συγκήτρια θα, θα αναφέρει σχετικά με την οδηγία των υπηρεσιών. Πρόεδρος, καλό ξεκίνημα. And uh, our will be back. Ε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα, γιατί είμαστε υπεύθυνοι και για τα δύο και είμαστε και για τα προσόντα. Χαιρόμαστε που υιοθετείτε τέτοια στιβαρή προσέγγιση Λοιπόν, να κάνουμε τη συζήτηση και στο τέλος του πρώτου γύρου θα μιλήσει η κυρία Κοράτσα Μπίλτ να μας πει πώς θα προσεγγίσει το θέμα στην ε, έκθεσή της. Έχουμε την κυρία Ράπτη εδώ που είναι σκιώδης για την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, από τους Φιλελευθέρους ο κύριος Μάντος, ο κύριος Ρούντες από τους Πράσινους, εγώ είμαι ο σκιώδης της ομάδας μου από το Ιγκούε δεν είναι κανείς αυτή τη στιγμή. Θα δούμε αν θα έρθει κανένας και κάποιος άλλος, όποιος ε, όλοι ευπρόσδεκτοι. Κυρία Ράπτη, έχετε το λόγο πρώτη. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και θα συμφωνήσω μαζί σας σε σχέση με αυτό που είπατε. Καλή αρχή. Νομίζω ότι κάναμε μια εξαιρετική αρχή. Η, τα όσα ανέπτυξε η εκπρόσωπος της Κομισιόν ε, με κάνουν να είμαι αισιόδοξη για τη δουλειά μας και για το αποτέλεσμά της. Ε, μας έδωσε αρκετές α, λεπτομέρειες, θα έλεγα πολύ περισσότερες από όσες τουλάχιστον εγώ περίμενα. Ε, αισθάνομαι ότι η εισήγηση της Κομισιόν είναι φιλόδοξη αλλά ταυτοχρόνως αισθάνομαι ότι έχει και στοιχεία ρεαλισμού. Με άλλα λόγια, αισθάνομαι πραγματικά ότι έχει στο μυαλό της τους Ευρωπαίους πολίτες με όλες τις ιδιότητες που αυτοί έχουν. Είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι καταναλωτές. Α, ασφαλώς χρειαζόμαστε χρόνο για να δούμε τις λεπτές εκείνες εκφράσεις και εκφάνσεις όλης της εισήγησης για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε και εμείς στο να δημιουργηθεί το καλύτερο δυνατό νομοθετικό πλαίσιο που να μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, θα εκφραστώ πάρα πολύ θετικά και για την πολύ καλή συνάδελφο, την κυρία Κοράτσα Μπίλτ, της οποίας η δουλειά μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ εδώ και τρία χρόνια σε αυτή την Επιτροπή. Ε, χαίρομαι που είναι εδώ άνθρωποι τους οποίους αφορά κυρίως η υπόθεση αυτή της ενίας αγοράς, όπως είναι οι επισκέπτες μας και νομίζω ότι και αυτοί, παρακολουθώντας τη συνεδρίασή μας και μιλώντας μετά με την Κοράτσα, θα μπορούν να συμβάλλουν στην δουλειά που κάνουμε εδώ. Ε, μερικά σημεία πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι μια πρώτη κουβέντα σήμερα. Ε, το πρώτο είναι και το υπογραμμίζω πάλι, καλωσορίζω την διάθεση και την ανακοίνωση της Επιτροπής θεωρώ θετικό ότι πραγματικά γίνεται πρακτικά μια πρώτη εκτίμηση για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η οδηγία στα κράτη-μέλη. Θεωρώ θετικό ότι έχουμε στο μυαλό μας μια περισσότερο αυστηρή λογική στην παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας, αλλά εδώ θέλω να βάλω ένα πρώτο αστερίσκο. Ε, να μην έχουμε στο μυαλό μας μόνο την τιμωρία, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο δεν βοηθάμε να πάμε μπροστά. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και το να παρέχουμε κάθε δυνατή τεχνική βοήθεια σε, ε, στα κράτη-μέλη, κυρίως στα κράτη-μέλη εκείνα που δεν έχουν προχωρήσει πολύ και παράλληλα να βοηθήσουμε στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Ε, θεωρώ εξαιρετικά θετικό το να υπάρχει συνεργασία με τους εθνικούς ε, φορείς και να προωθηθούν συγκεκριμένες δράσεις που θα διασφαλίζουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες όλων των Ευρωπαίων πολιτών ανεξάρτητα από εθνικότητα, ανεξάρτητα από τόπο διαμονής. Ε, η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και κανόνων, το είπε και η κυρία Κοράτσα, είναι ένα θέμα που θέλει πολλή συζήτηση και θέλει και ένα χειρισμό. Γιατί κάθε κράτος μέλος έχει τις ιδιαιτερότητές του και κάποια προχωρούν πιο γρήγορα, κάποια λιγότερο γρήγορα. Εκεί νομίζω ότι πρέπει όλοι να κάνουμε προσπάθειες ώστε να υπάρξει ένας γοργός βηματισμός. Ο γοργός αυτός, ο γρήγορος αυτός βηματισμός δεν θα πρέπει όμως να, είναι, ε, να έρχεται κόντρα στην προστασία του καταναλωτή. Για μας είναι πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα το θέμα της προστασίας του καταναλωτή. Υπέρ του καταναλωτή όμως θεωρούμε ότι θα είναι σαφώς η σωστή λειτουργία των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης και βέβαια το να μπούμε στην καινούρια εποχή με τα κέντρα δεύτερης γενιάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ε, πραγματικά προσβλέπουμε πολύ σε αυτήν την ε, σε αυτά τα κέντρα δεύτερης γενιάς. Δεν θέλω να προχωρήσω παραπάνω. Ε, τελειώνω εκφράζοντας και πάλι την αισιοδοξία μου σε σχέση με όλη αυτή τη δουλειά που ξεκινάμε σήμερα και να πω ότι είμαι στη διάθεση ε, της εισηγήτριας μαζί με τους εξαιρετικούς συναδέλφους Κιώδης να δουλέψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάντερς. Ευχαριστώ. Αντικαθιστώ και όλοι. ο οποίο συμφωνεί με τα συμπεράσματα της ανακοίνωσης, προσθέτει κάποια. Η Κομισιόν εισαγωγικά λέει ότι ε, συμφωνεί με τις παρατηρήσεις αυτές, δεν θα τις διαβάσω. Τώρα, το έλλειμμα στη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία δεν αφορά μόνο αυτή την νομοθεσία, αυτή την οδηγία. Ε, ίσως θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε κανονισμό. Χαίρομαι γιατί μετά το ΕΛΚ μετά από κάποια χρόνια έχει πιστεί κανονισμοί αντί οδηγίες. Γιατί τι συμβαίνει πάντα. Η μεταφορά των οδηγιών δημιουργεί πρόβλημα. Χρειάζεται ολόκληρη οργάνωση δηλαδή για να αξιολογήσει αν έγινε σωστά. Γιατί να μην αρχίσουμε πιο απλά να εφαρμοστεί κανονισμός ή δυνατόν. Εγώ θέλω να κάνω αυτή την πρόταση. Ο κύριος Λόγκεγκαρτ χαίρεται επίσης ε, γιατί φαίνεται ότι το έλλειμμα ε, βελτιώνεται. Κλείνει λίγο το κενό, αλλά όχι αρκετά, σε ό,τι αφορά τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία. Και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που χάνουμε, με όλες τις καλές αναφορές που έχουμε, χάνουμε την ε, αναφορά στον κόσμο, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι κάνουμε. Επιμένω στην επικοινωνία. Σκεφτείτε πώς μπορεί να βελτιωθεί, ούτως ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να ξέρουν τι κάνουμε. Στο βαθμό που δεν ξέρουν τι κάνουμε, χάνουμε υποστήριξη για όλη την καλή μας τη δουλειά. Και αν δεν στηρίζουν οι πολίτες πια την Ευρώπη, πάει. Τότε η δουλειά μας χάνεται. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ. Ήμουν σύντομος. Και βέβαια υπάρχει εδώ υποστήριξη από το Σκιώδη στην Άννα Μαρία. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρούιλε. Χαίρομαι για την καλή συνεργασία πάλι με την κυρία Κοράτσα Μπίλντ. Θα περιμένω να δω τι θα προκύψει, δεν έχω πολλά σχόλια. Δεν θα παρεκτραπώ για να πω άλλα θέματα όπως το κάνει τόσο ωραία ο κύριος Μάντερς. Όχι, εγώ δεν θα τον ακολουθήσω. Οπότε σταματώ εδώ. Okay, um, Καλώς. Και από μένα κάποια σχόλια. γιατί θα είμαι σκιώδη σε αυτή τη σημαντική πρόταση. Μαζί με τον κύριο Μάντερ, μαζί με την κυρία Ρούλε, οι τρεις μας δουλέψαμε την αρχική πρόταση που ολοκληρώθηκε το 2006, οπότε είναι στο DNA μας αυτή την Επιτροπή. Τότε ήμουν σκιώδης της ομάδας ΕΛΚΑ Ευρωπαίοι Δημοκράτες για όλη την πρόταση και με απασχόλησε τέσσερα χρόνια η πρόταση αυτή στο σύνολό της. Κάποια γενική παρατήρηση θα κάνω. Γιατί καμιά φορά πιστεύουμε, πιστεύει ο κόσμος δηλαδή, ότι αυτό το κοινοβούλιο νομοθετεί με αποσυνδεδεμένο τρόπο, σαν να μην ε, ε, υπάρχει συνέχεια. Ε, σε μια θητεία δουλεύουμε και μετά δεν υπάρχει συνέχεια. Εμείς ε, αφιερώσαμε πάρα πολύ χρόνο και αυτό δείχνει ότι το κοινοβούλιο πολύ σε βάθος ε, συμμετέχει και φροντίζει για τη σωστή εφαρμογή. Και προκειμένου δουλέψαμε στενά και με την Κομισιόν. Το θέμα της ε, εφαρμογής στην εθνική νομοθεσία αυτής της οδηγίας ήταν ευρύτερη από ότι η εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης οδηγίας στην ενιαία αγορά. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι το έργο αυτής της Επιτροπής από το 2009 και που θα συνεχίσει και στις δημόσιες συμβάσεις θα παρακολουθούμε και αυτά. Γιατί στο μέλλον θα έχουμε λιγότερα νομοθετήματα. Θα παρακολουθούμε όμως αυτά που ήδη έχουμε θεσπίσει. Αυτό είναι σαφής ένδειξη με βάση την έκθεση. Αυτά τώρα για την ιστορία, το ιστορικό σε αυτά τα πλαίσια η έκθεση πρέπει να είναι μια αυστηρή, μια στιβαρή έκθεση η κυρία Κοράτσα Μπίλντ είπε ότι αγανακτεί για το γεγονός ότι οι αρχικές φιλοδοξίες από την οδηγία που βρήκαν σύμφωνες όλες τις πολιτικές, όλα τα πολιτικά κόμματα και, οι, ε, και τις, κάποιες κυβερνήσεις δεν ε, υλοποιούνται και αυτό δεν είναι αποδεκτό. Όλοι ευθυνόμαστε στα πλαίσια της ε, πράξης για την ενιαία αγορά που την παρακολουθήσαμε, παρακολουθήσαμε ε, ε, έπρεπε να εφαρμοστεί ένα πολιτικό πρόγραμμα, όχι μόνο νομοθετικό. Και πολλές πτυχές της πράξης για την ενιαία αγορά επικεντρώνονται στην εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Παράλληλα, έχουμε και την έκθεση του Άντριου Σβάμπ για το πώς θα είναι υπόλογα τα κρατημέλη αν δεν ανταποκρίνονται και δεν παρέχουν ε, οικονομικά ωφέλη και αν δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας για τους πολίτες μαζί με βιώσιμη ανάπτυξη, με δημιουργία θέσεων εργασίας. Και δεν το λέω γιατί είναι υπέρμαχος όλων αυτών μεγάλο, η κυρία Ρούλε. Όλοι τα πιστεύουμε αυτά. Όλα αυτά πρέπει να παραδοθούν, αλλιώς θα κάνουμε βήματα προς τα πίσω ή θα παραμείνουμε στάσιμοι. Οι ανακοινώσει τη Κομισιόν λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Τι θα κάνουμε λοιπόν εν προκειμένου. Πρώτα απ' όλα νομίζω και είναι πολύ καλό που έχουμε και επιχειρηματικό ακροατήριο από μια χώρα που μάλλον ε, συμμορφούνται σε περισσότερο με την οδηγία για τις υπηρεσίες από άλλη. Τα δεδομένα θα το αποδείξουν αυτό. Λοιπόν, χρειαζόμαστε επιχειρήσεις που θα πρέπει να ενίστανται σε ενώπιόν μας πολύ περισσότερο, γιατί Μέρος του προβλήματος με τις υπηρεσίες από αυτά που εντοπίστηκαν είναι τα κρυφά εμπόδια που ήταν κρυμμένα στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών. Ε, διακριτικά εμπόδια που δημιουργούν διακρίσεις. Ε, ακούσαμε για κάποια που υπάρχουν και τώρα αυτά αναφέρονται ξεκάθαρα στην έκθεση. Πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όροι, προαπαιτούμενα. για να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που εξακολουθούν να ορθώνονται. Ε, δεν μπορούν οι εταιρείε ε, να παράσχουν υπηρεσίες γιατί δεν τηρούν κάποιες νομικές προϋποθέσεις και διατάξεις, ε, υποχρεώσεις ασφάλισης κλπ. κλπ. Πολλά άλλα ακόμα. Αυτά εντοπίστηκαν σε μια μελέτη από το 2002 και το 2003. Μέρος του προβλήματος που εντοπίστηκε ήταν ότι οι επιχειρήσεις που προσπαθούν να συσταθούν αποθαρρύνονται τόσο πολύ από όλες αυτές τις νομοθεσίες που έκαναν κάτι άλλο. Φαντάζομαι ότι εξακολουθεί να σημαίνει αυτό, απλώς δεν το ξέρουμε επαρκώς. Και θέλουμε οι επιχειρηματικές οργανώσεις να μας βοηθήσουν για να εντοπίσουμε τα εμπόδια που υπάρχουν. Τα άρθρα 15 και 16 στην Οδηγία για τις Υπηρεσίες και η βασική ρήτρα για την ε, ελευθερία παροχής υπηρεσιών ήταν η πιο δύσκολη συμβιβαστική λύση που άνοιξε τις ευκαιρίες. Αυτή ήταν η συμβιβαστική λύση κλειδί που ξεκαθάρισε ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν ε, υποχρεώσεις σε κάποιον που θέλει να παράσχει υπηρεσίες προσωρινά ή μόνιμα. Αυτό είναι η καρδιά της πρότασης παροχή υπηρεσιών. Στην έκθεσή μας και το λέω στην εισηγήτρια, πρέπει να επικεντρωθούμε με βλέμμα οξύτατο θα έλεγα στην πρόταση αυτή. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό δεν θα δοθεί συνέχεια σε τίποτα άλλο. Αν τα κράτη-μέλη συνεχίσουν να διατηρούν τους περιορισμούς θα έχουμε σαφώς αποτύχει ε, με αυτή τη φιλόδοξη οδηγία υπηρεσιών. Σας το λέω αυτό έτσι ομά. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό με μεγάλη ένταση. Και ως μέλος της ακρόασης πρέπει να καλέσουμε την Κομισιόν να μας βοηθήσει με, και να έρθουν κάποια κράτη-μέλη επίσης που δεν προχωρούν θέλουμε και αξιωματούχους και υπουργού από κάποια κράτη-μέλη να έρθουν να μας εξηγήσουν γιατί δεν συμμορφούνται με τις προϋποθέσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε εξουσίες να τους αναγκάσουμε να έρθουν, αλλά πολλοί από τους συναδέλφους από τις χώρες που δεν ε, είναι καλοί μαθητές, πρέπει να έρθουν και να μας εξηγήσουν τι δεν πάει καλά. Να δούμε τους στόχους, γιατί το κάνουν. Δηλαδή πιστεύουν ότι ο προστατευτισμός είναι η απάντηση στα σημερινά μας προβλήματα. Αυτό είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση, η ενημέρωση. Και κάτι άλλο που νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε δεν είναι τόσο η ύπαρξη ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης, αλλά γιατί οι επιχειρήσεις δεν τα γνωρίζουν αυτά τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης. Ένα μέρος του θέματος γύρω από την οδηγία για τις υπηρεσίες ήταν να δίδονται πηγές ενημέρωσης. Και μάλιστα τα κράτη-μέλη που επένδυσαν πολύ χρόνο, χρήμα, πόρους για να δημιουργήσουν αυτά τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης και πολλά μάλιστα είναι πολύ ευραία και δουλεύουν εξαιρετικά και καμιά φορά είναι και ευρύτατα, πολύ συνεκτικά. Επιτρέπουν σε έναν πάροχο που πρέπει να καταχωριστεί γιατί έχει ιδιαίτερη μια ειδική κατηγορία επιχειρήσει, δηλαδή εφοδιασμός με τρόφιμα, ασφάλεια τροφίμων, και μπορούν να πάνε και να καταχωριστούν στην αρμόδια αρχή. Αυτό έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλιώ μόνο θεωρητικολογού όταν μιλάμε για αυτά τα προαπαιτούμενα. Αυτό επίση που πρέπει να δούμε είναι τα κράτη-μέλη που επένδυσαν πολύ στα κέντρα ενιαία εξυπηρέτηση ε, να μας πούν πόσο λίγες επιχειρήσεις τα γνωρίζουν. Και κάτι άλλο που πρέπει επίση να εξετάσουμε είναι το χαμηλό επίπεδο ευαισθητοποίηση για τις δυνατότητες ενημέρωσης που υπάρχουν για τις επιχειρήσεις που θέλουν να εγκατασταθούν σε μια άλλη χώρα. Γιατί είναι σαν μια επιχείρηση να επενδύσει ένα μεγάλο καινούριο ωραίο προϊόν, ξεχνώντας όμως να ενημερώσει ότι υπάρχει το προϊόν. Αυτή είναι η αποτυχία των κρατών μελών. Και επειδή δεν υπάρχει εσωτερικό, δεν υπάρχει εσωτερικό κίνητρο ε, για την ε, κοινοποίηση της ενημέρωσης. Πάντως, ε, πολλές επιχειρήσεις μπορούν να μας βοηθήσουν και ίσως θα πρέπει να καλέσουμε και τον αρμόδιο επίτροπο να μας στηρίξει με τον προϋπολογισμό έρευνας που έχουμε ε, και μπορεί να μας βοηθήσει εδώ. Επίσης κάτι άλλο, κάτι άλλο που αφορά την προηγούμενη δουλειά μας. Νομίζω ότι Πρέπει να αναφερθούμε στα θέματα αμοιβαία αναγνώριση προσόντων και αυτό είναι κομμάτι τη ευθύνη μα. Επίση, τα πρότυπα, ένα άλλο τομέα. Συμφωνήσαμε ότι ε, είναι πολύ σημαντικό το πακέτο των προτύπων που για πρώτη φορά ε, περιλαμβάνει την δυνατότητα για την Κομισιόν να ε, αναθέσει την κατάρτιση στάνταρ για τις υπηρεσίες και υπάρχει αυξανόμενη δραστηριότητα από τους καταναλωτές που θέλουν να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες διασυνοριακά με, και να ε, υπάρχουν κάποια σημεία αναφορά σε συγκριτική αξιολόγηση και πρότυπα για τις υπηρεσίες. Υπάρχει συγκεκριμένο προαπαιτούμενο στην Οδηγία Υπηρεσιών για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και αναβάθμισης προτύπων για τις υπηρεσίες. Θα Θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν, γιατί αυτό είχε αναφερθεί στην έκθεση. Τα κράτη-μέλη έχω την εντύπωση ότι αγνόησαν αυτό το κομμάτι. Το αγνόησαν μέχρι τώρα, γιατί ε, είχαμε το, τη συνοδευτική νομοθεσία για τα πρότυπα, το companion, αλλά ε, τώρα πρέπει να το κοιτάξουμε ανεξάρτητα το θέμα, γιατί θα διευκολύνει τις διασυνοριακές υπηρεσίες και αυτά που είπαμε για τα πρότυπα θα ξαναμπούν σε τροχιά και θα ισχύσουν. Θα υπάρξει δηλαδή μια έκθεση ενημέρωσης τους επόμενους 18 ε, μήνες μέχρι τις εκλογές ε, για να ε, ολοκληρώσουμε το νομοθετικό έργο αυτής της Επιτροπής. Αυτά είχα να πω για την έκθεση. Νομίζω ότι η συγκίτρια θα πρέπει να κάνει διαβουλεύσεις με όλες τις πολιτικές ομάδες και τους ε, συντονιστές για να σχεδιάσει τη συνέχεια που θα δοθεί και πώς θα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ακρόαση. Ε, μακρηγόρησα λίγο ως κοιόδης και ως πρόεδρος, αλλά έχουμε χρόνο πολύ για τη συζήτηση αυτή. Οπότε έδωσα, τον εαυτό μου στη, έδωσα στον εαυτό μου την πολυτέλεια να μακρηγορήσω. Δεν θα το έκανα αλλιώς. Ε, ευχαριστώ πολύ. Τώρα άλλοι συνάδελφοι. ο κύριος Μπαλτασάρε, Μπαλτασάρε, ο κύριος... Σας έπεισα μου φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ Μάλκομ. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα το απόγευμα θεωρώ ότι είναι περίοδος περισυλλογής, διότι είναι ελάχιστοι συνάδελφοι που έμειναν εδώ να ακούσουν την έκθεση της κυρίας Ανάς Μαρίας Κορατσαμπίλτ ακούστηκαν κάποιες ε, σκέψεις ε, οι οποίες πηγαίνουν πολύ περισσότερο από την έκθεση αυτή αυτή και έχουν σχέση με τις εργασίες μας και το τι κάνουμε εμείς εδώ στην Επιτροπή μας. Πολλές φορές θα θέλαμε να πάμε πολύ πιο πέρα και θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι θέμα επικοινωνίας, διότι όλοι είμαστε πεπισμένοι ότι εν περίοδο κρίσης ε, η εσωτερική αγορά αποτελεί τη λύση. Αυτή λοιπόν η εσωτερική αγορά έχει μεν κάποια ωφέλη, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει και κάποια δικαιώματα για τους καταναλωτές, ώστε να θεωρούν αυτούς ασφαλείς και να ε, τιμούν το όνομα της Επιτροπής μας. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση, να δούμε κατά πόσον πρόκειται για οδηγία ή για κανονισμό, διότι το να λέμε ότι πρέπει να τηρούνται και να δεσμεύονται ε, τα, τα κράτη-μέλη ότι θα τηρήσουν τα όσα προβλέπει είναι πολύ σημαντικό. Ε, δεν ξέρω αν η χώρα μου περιλαμβάνεται μέσα ε, σε αυτές τις χώρες που τηρούν ή δεν τηρούν την οδηγία. Καλό θα ήταν να κατονομάσουμε όλους όσους δεν τηρούν ε, την οδηγία, αν πραγματικά θέλουμε να πάμε έτσι περιπέτερο και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Δεδομένης λοιπόν και της συγκεκριμένης συγκυρίας και και τη ώρα και το γεγονός ότι, το γεγονός ότι είναι ελάχιστοι συνάδελφοι που είναι εδώ και έχουμε απλώ του τους προσκεκλημένους εδώ, Καλό θα ήταν λοιπόν να γνωρίζετε ότι οι εργασίες της Επιτροπής μας ε, οδηγούν σε αποτελέσματα τα οποία πηγαίνουν πολύ πιο πέρα από ε, τα ωφέλη για τους λίγους. Πηγαίνουμε πολύ πιο πέρα γιατί θέλουμε να έχουμε ωφέλη και να έχουμε μια πολύ πιο ασφαλή αγορά στην Ευρώπη, από την οποία να μπορούμε να αποφεληθούμε όλοι. Σε ευχαριστώ πολύ, ε, Μάλκολμ, που μου έδωσε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή σας. Νομίζω ότι ίσως η κυρία Φρονσουά Κονσέ θα μπορούσε να μας πει, να μας απαντήσει μετά από τα όσα άκουσε και μετά θα δώσω πάλι το λόγο στην κυρία να μας πει ορισμένε ιδέες σχετικά με το να προχωρήσουμε. uh, πρώτα απ' όλα θα απαντήσω στο ερώτημά σας για τα πρότυπα. Όπως γνωρίζετε, ξεκινήσαμε ήδη να δουλεύουμε το θέμα των προτύπων και στείλαμε με εντολή για οριζόντια πρότυπα, αλλά το ξεκινήσαμε αυτό και συνεργαζόμαστε με την ΣΕΝ, με την, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης και με σκοπό να εκπονήσουμε πρότυπα και να βρούμε πιθανόν οριζόντια ε, οριζόντια πρότυπα της υπηρεσία. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Οπωσδήποτε χαιρετίζουμε την υποστήριξη Επιτροπής σας για τη δουλειά που κάνουμε. Δεν είναι εύκολο το έργο μας και θα ήθελα να αναφέρω ένα πράγμα το οποίο είναι σημαντικό. Κανένα κράτος μέλος μόνο του μεμονωμένα δεν θα μπει στη μαύρη λίστα. Απλά και μόνο η δυσκολία είναι ότι υπάρχει ποικιλότητα διαφορ... κανόνων, διαφορετικές νομοθεσίες και το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένε απαιτήσει νομικής μορφής. Ε, τα κράτη έχουν κάποια περιθώρια, κάποια διακριτική ευχαίρεια, αν θέλετε, όσον αφορά την αναλογικότητα και την εκτίμηση της αναλογικότητας. Και είναι δύσκολο να τα ενοποιήσουμε όλα αν θέλετε, να τα σαρώσουμε. Άλλωστε ε, σημαντική θα είναι αυτή η μελέτη των νομοτήμων, διότι δεν μπορεί κανείς να δοκιμάσει την αναλογικότητα πάντοτε, πρέπει να τη δούμε σχετικά, να συγκρίνουμε το ένα σύστημα με το άλλο. Το γεγονός παραμένει όμως ότι η σημασία που μπορεί να δοθεί από πολιτικής απόψεως σε θέματα όπως αυτό θα μας βοηθήσει διότι έτσι κι αλλιώ αυτό το έργο θα πάρει πολύ χρόνο. Ε, σχεδόν το, το κάθε επάγγελμα έχει να κάνει με ορισμένους προδιαγραφέρμους απαιτήσει ε, νομικής φύσεως και σε σχέση με τους μετόχους των επιχειρήσεων. Όσον αφορά τις πληροφορίες, την ενημέρωση, ναι, αυτό ε, είναι ένα από τα θέματα οι επιχειρηματικές οργανώσεις συμφωνούν με αυτά τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης και είναι διατεθειμένες να μας βοηθήσουν επιχειρήσεις. Η Business Europe ε, φτιάχνει αρκετές εκθέσεις, καταρτίζει εκθέσεις και μας ακολουθούν, ε, συμφωνούν με τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης. Ε, αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι σε εθνικό επίπεδο να είναι ενημερωμένο ο κόσμος μπορεί αυτά που λέμε εδώ να μην γίνουν γνωστά όσο θα θέλαμε ε, στις διάφορες χώρες. Συνεπώς, πραγματικά, αυτά τα κέντρα μιας εξυπηρέτησης μπορούν να βοηθήσουν και προτού τα καταστήσουμε αρκετά γνωστά, ε, επειδή γνωρίζουμε πώς ε, τον κίνδυνο που ενέχει η δημοσιότητα που μπορεί κανείς να δώσει σε κάτι. επιθυμούμε πράγματι να δώσει συνέχεια στην ανακοίνωσή μας η Επιτροπή και εμεί θα παρακολουθήσουμε ε, τις εργασίες σας με, ε, με δραστήριο τρόπο με όλα τα κράτη-μέλη. Ήδη ξεκινήσαμε και αυτό θα το συνεχίσουμε τα επόμενα δύο χρόνια. Ευχαριστώ. Good, thank you very much. Um, Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα τον τελευταίο λόγο στην εισηγητριά μας σχετικά με τα μελλοντικά βήματα. Πρόεδρε, χαιρετίζω πολύ αυτή τη συζήτηση που έγινε, που καταδεικνύει ότι έχω μια ισχυρή εντολή, δηλαδή να φτιάξω μια ισχυρή σημαντική έκθεση με την υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων εδώ και αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με ε, την έκθεσή μου. Στους συναδέλφους από τους σοσιαλιστές εκτιμώ το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και ότι έχουμε την ίδια αυστηρή προσέγγιση σχετικά με την υλοποίηση και όχι μόνον όσον αφορά τις ε, κυρώσεις αλλά και τεχνική υποστήριξη. Αυτό μου επιτρέπει να υπογραμμίσω τη σημασία που έχει η ανταλλαγή των καλών πρακτικών και της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών σχετικά με αυτά που πρέπει να εφαρμόσουμε και πώς μπορούμε να μάθουμε από αυτά. Η συνεργασία μεταξύ εθνικών οργανισμών είναι πολύ σημαντική. Παράλληλα, θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που η Επιτροπή άρχισε ε, να εφαρμόζει διαδικασίες πριν από τις παραβιάσεις. Δεν πρέπει να μας φοβίζουν. Αποτελούν μέρος της νομοθεσίας και δεν είναι κάτι ότι, για το οποίο πρέπει να ντρέπεται κανείς, αλλά αυτό γίνεται για το καλό των Ευρωπαίων πολιτών για να προωθήσουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία τα κράτη-μέλη δεν θα αντιμετώπιζαν την κρίση που αντιμετώπιζαν τώρα αν είχαν εφαρμόσει την νομοθεσία που υπάρχει. Συνεπώς πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να υπάρχει όταν ε, τα, τα, κράτη, τα κράτη δεν έχουν περιθώρια λιγμών. Και χαίρομαι που αυτό ακολουθεί η Κομισιόν. Αυτό πρέπει να γίνει ε, σε διάλογο με τα κράτη-μέλη και χαιρετίζω την πρότασή σας Μάλκομ να έχουμε μία ακρόαση με την ε, παρουσία των κρατών μελών και να μας πούν τι πιστεύουν, πώς αυτός ο κατακαιρματισμός ε, της, με, ε, της μεταφράσης των πρακτικών, πώς μεταφράσει στην πράξη και τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα. Αυτό που κάνει η Επιτροπή είναι πολύ καλό και πρέπει να ακολουθήσουμε τα βήματά της. Τώρα, ε, τι πρέπει να κάνουμε για να φροντίσουμε την προστασία των καταναλωτών. Πάλι από του σοσιαλιστέ μα το είπαν. Γι' αυτό το λόγο η πλήρη εφαρμογή του άρθρου 20 για τη μη διάκριση είναι τόσο σημαντική. Και θα πρέπει να προχωρήσουμε και εδώ. για να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες, να υπάρξει λιγότερη σύγχυση, να υπάρχουν σαφέστεροι κανόνες για τους καταναλωτές. Ε, συνάδελφο από το Άλντε οι κανονισμοί μας ε, ε, εντάσσονται σε αυτήν την ομάδα. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω εδώ κύριε Πρόεδρε είναι ότι θα χρησιμοποιήσω οτιδήποτε μας προσφέρει αυτή η οδηγία για να ξεπεράσουμε αυτό το πνεύμα, να μην ε, ξεκινήσουμε μια νέα νομοθετική διαδικασία για να ενημερώσουμε, να επικαιροποιήσουμε αυτή την οδηγία. Αυτή τη στιγμή έχουμε νέες έννοιες των υπηρεσιών. Δηλαδή πουλάμε αγαθά και υπηρεσίες μαζί, ε, πουλάμε λύσεις πακέτα. Είναι ένα μείγμα, πουλάμε ένα πακέτο με πολλά προϊόντα, αν θέλετε, και πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες εξελίξεις, διότι οι πάροχοι υπηρεσιών συνέχεια επικαιροποιούν, ενημερώνουν τις υπηρεσίες τους ε, από το 2006 μέχρι σήμερα. Και πρέπει να προσαρμοστούμε στο γεγονός ότι ο, κινη, ο κόσμος, ο κινητός κόσμος αν θέλετε, δεν υπήρχε. Ε, μια ολόκληρη γενεά χρησιμοποιεί υπηρεσίες ε, με κινητά μέσα, δηλαδή με την κινητή τηλεφωνία. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη ε, στην εφαρμογή των μέτρων μας. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, η ανακοίνωση, το είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, το, αυτά τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να ανταποκριθούμε στην ανάγκη της επιχειρηματικής κοινότητας να χρησιμοποιήσει σωστά την ενιαία αγορά και να παρέχει ε, ε στους υπηκόους των κρατών μελών αυτές τις πληροφορίες. Προσπαθώ να καλύψω όλους το γεγονός ότι υπάρχει υποστήριξη όλων των, του πολιτικού φάσματος. ευχαριστώ, Πρόεδρε, που είπατε ότι η οδηγία υπηρεσιών δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως. Συμφωνώ. Ελπίζω ότι θα φτιάξουν ένα πακέτο το οποίο θα πείσει τα κρατημέλη ότι σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται ανάμεσα ε, στη λιτότητα και την ανάπτυξη, το γεγονός ότι δεν έχουμε πραγματική ελεύθερη διακίνηση των υπηρεσιών είναι κάτι το οποίο δεν έχει συνοχή και θα πρέπει να το διασυνδέσουμε ε, με την ατζέντα για την ανάπτυξη και θα πρέπει κάτι να, προσ... να συνεισφέρουμε ε, στη συνάντηση κορυφής του Δεκεμβρίου. Να εξηγήσουμε τι θα είναι αυτή η ενιαία αγορά. Η ατζέντα ε, αφορά την επόμενη χρονιά, δηλαδή μέχρι το φθινόπωρο του χρόνου θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες μας και θα υπάρχει την άνοιξη μια ακρόαση και προσβλέπω να συνεργαστώ με τους ενδιαφερόμενους, με τους παίκτες του επιχειρηματικού κόσμου, ώστε να λειτουργήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you very much. Ε, ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Και νομίζω ότι αν έπρεπε να είναι κάποιος συζητητής για το θέμα αυτό, ε, σίγουρα είστε εσείς. Προσωρινά τώρα να σας πω ότι είχαμε σκεφτεί να υπάρχει μια ακρόαση, ένα εργαστήριο το Φεβρουάριο και από εκεί και πέρα ε, μέχρι τις 15 Μαρτίου θα λάβετε και τις μεταφράσεις και από εκεί και πέρα θα προχωρήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας. Ε, ελπίζω να υπάρξει και ένας γύρος τραπέζης με τους κοιόδης εισηγητές. Ε, δεν ξέρω και αν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συναντηθούμε. Θα περιμένουμε να ακούσουμε αν υπάρξουν κάποιες περαιτέρω εξελίξεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα. Και Μπορεί να θελήσετε να συμπεριλάβετε και όλα αυτά στη μελέτη σας. Είναι πολύ σημαντικό ε, να τονίσουμε ότι πριν από ακριβώς έξι χρόνια ψηφίσαμε στην Ολομέλεια για την οδηγία για τις υπηρεσίες, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Πέρασε αρκετό καιρό έκτοτε το Κοινοβούλιο έκλεισε το ζήτημα και ξέρω ότι η κυρία Γκέπχορτ, η οποία δυστυχώς δεν είναι εδώ σήμερα, αλλά ήταν τότε η συγγήτρια, θα συμφωνεί σίγουρα μαζί μας και θα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και αυτή για την έκθεση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τη συζήτηση. Το θέμα ολοκληρώθηκε τώρα και το επόμενο σημείο είναι η έκθεση του κυρίου Μπαλτασάρε για το πρόγραμμα δράσης για τα ταελωνία έχουμε λίγο χρόνο και αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν είναι εδώ ούτε σκιώδεις συζητητές. Ε, λείπει και ο κύριος Κοφεράτη σίγουρα. Δεν ξέρω αν είναι και κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, η Κομισιόν είναι εδώ. Αυτό είναι καλό. Να ζητήσουμε λοιπόν από τους σοσιαλιστές ε, να πούνε στον κύριο Κοφεράτη να έρθει το συντομότερο δυνατόν και μετά να συνεχίσουμε. Ο κύριος Μπαλτεσάρο είναι παρόν και έτοιμος να μιλήσει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος από τη γραμματεία των σοσιαλιστών. No. Sono andati tutti via con ah. Tarabella. Έφυγαν όλοι με τον Ταραμπέλα, λέει ο κύριος Μπαλτασάρε. Θα παραδώσω την προεδρία στην ε, ε, αντιπρόεδρο, στην κυρία Βανίλ. Θα πάρει τη θέση μου και μετά θα δώσουμε τον το λόγο στον κύριο Μπαλτασάρε. Sì, grazie Presidente. Io sarò molto breve. Μισό λεπτό να αναλάβει καθήκοντα Πρόεδρος. And she is in charge. Undisputably in charge. Και μετά θα κάνει κουμάντα αυτή. Merci. Alors je mette la traduction. Alors la traduction. Ok. Voilà. Ωραία, θα είμαι πολύ σύντομο, λέει ο κύριος Μπαλτασάρε. Αυτό το σχέδιο έκθεση ε, προσπαθεί να επιτύχει τους εξής στόχους. Για λόγους προβολής και νομικής αφήνειας, ελπίζω οι προτεραιότητες να μεταφραστούν σε συγκεκριμένους στόχους. Αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 6, τροπολογία 14, και ελπίζω να συμπεριληφθούν όλα αυτά στο διατακτικό του κανονισμού. Πάντα για το άρθρο 6 θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ενδεκτική αναφορά του προπολογισμού που μας ε, επιτρέπει να κάνουμε και προσθήκες για τεχνικές δαπάνες και ε, τροποποίησεις υπό την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 2. Επίσης ε, λαμβάνονται υπόψη και το θέμα της χρηματοδότησης, εν αναμονή ε, της ε, απόφασης για τις πολυετής δημοσιονομικές προοπτικές, ελπίζω να ολοκληρωθούν με αίσιο τέλος. Ε, λαμβάνονται υπόψη και θέματα συντήρησης των ε, συστημάτων πληροφορικής, ε, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους βάσει του προϋπολογισμού του προηγούμενου ε, προγράμματος ε, Τελωνία 2012, διότι μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού δίνεται για το θέμα αυτό. Για να λάβουμε υπόψη τις διάφορες δράσεις των τελωνιακών αρχών, πρέπει το πρόγραμμα να καλύπτει και τις κοινέ δράσεις, ε, την ανάπτυξη των δυνατοτήτων πληροφορικής, του ανθρωπίνου δυναμικού επίσης, αλλά πρέπει να καλύπτει και τις τεχνικές δυνατότητες ε, όλης ε, αυτής της διαδικασίας. Και τέλος, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ε, εναρμόνιση και τυποποίηση των τελωνιακών διαδικασιών. Αυτή λοιπόν ήταν η τοποθέτησή μου. Κάποιοι συνάδελφοι παρουσίασαν πάνω από 40 τροπολογίες, κυρίως η κύριοι Κοφεράτη, Γκρέντς, η κυρία Λεγκρίπ, η κυρία Βαλντεν Κάρμερ. Μετά από αναλυτική εξέταση των προτάσεων τροπολογίας μπορώ να σας πω ότι συμφωνώ με τη μεγάλη πλειοψηφία των τροπολογιών που κατατέθησαν, ιδίως ε, αυτές του κυρίου Κοφεράτη και του κυρίου Σμιτ οι οποίοι κύριοι Κοφεράτη και Σμιτ προτείνουν, όπως ακριβώς λέει η έκθεσή μου, το άρθρο 5 να περιορίζεται μόνο στη διευκρίνηση των γενικών στόχων και να ε, περάσουμε στους ειδικούς στόχους στο επόμενο άρθρο, δηλαδή στο άρθρο 6, το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερο να μιλάμε για συγκεκριμένους στόχους και όχι για προτεραιότητες. Και θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι όσον αφορά τις προτάσεις τροπολογίας που ε, ε, κατέθεσε η κυρία Λεγκρίπ, συμφωνώ προς το περιεχόμενο, παρά το γεγονός ότι δεν εγκρίνω τη διαφορετική διατύπωση που μου προτείνει. Ε, νομίζω ότι στο τέλος όμως με κάποιους συμβιβασμούς θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Τη μόνη αρνητική στάση την έχω για τις ε, ε, τροπολογίες της κυρίας Βάντερ Κάμελ, κυρίως τις τροπολογίες 45 και 46 που είναι αντίθετη στο άνοιγμα του προγράμματος σε χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία προσχώρησης και θεωρώ ότι η στάση αυτή είναι λανθασμένη, διότι δεν συνάδει και με τα όσα προβλέπει η συνθήκη και επίσης γιατί ως ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουμε ένα τεολωνιακό σύστημα το οποίο να είναι αποτελεσματικό, να είναι ε, διασυνδεδεμένο και να υπάρχουν και κατάλληλες υποδομές, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και χώρες με τις οποίες έχουμε σχέσεις ως Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε γιατί είναι γειτονικέ χώρες, είτε γιατί βρίσκονται καθοδόν προς προσχώρηση ή γιατί υπάρχει εταιρική σχέση. Ε, Υπάρχουν στενές λοιπόν σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό καλό θα ήταν να υπάρχουν τελωνιακοί ε, κώδικες που να είναι όσο το δυνατόν πιο ε, συγγενείς με αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να υποστηρίξουμε αυτές τις χώρες διότι ο ρόλος τους είναι συμπληρωματικός με το ρόλο που διαδραματίζουν τα τελωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω λοιπόν ότι με αυτές τις τροπολογίες θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ικανοποιητικό συμβιβασμό και να προχωρήσουμε από εκεί και πέρα, να εγκρίνουμε την έκθεση στις 18 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή Εστερικής Αγοράς και από εκεί και πέρα στο στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου θα περάσει από την Ολομέλεια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους για την αλληλεγγύη τους και την παρουσία τους, λέει ο κύριος Μπαλτασάρε. Ε, ευχαριστώ κύριε Μπαλτασάρε. Είμαστε ελάχιστοι εδώ στην αίθουσα. Ως πρόεδρος λοιπόν θα μιλήσω εγώ πρώτη και θα σας πω ότι συμφωνώ απολύτως για τις τροπολογίες 45 ε, και 46 και για να μην υπάρξουν και άλλοι ε, προβλήματα και για να υπάρχει και απαραίτητη ασφάλεια που ζητούν οι πολίτες πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις χώρες οι οποίες ε, είναι σε πορεία προσχώρησης και θα πρέπει να το τονίσουμε. Σας ευχαριστώ για τη δουλειά σας και να δώσω το λόγο στον κύριο Μάντερς διότι δυστυχώς νομίζω ότι οι υπόλοιποι σκιώδεις δεν έχουν έρθει. Κύριε Μάντερς έχετε το λόγο. And shadow actually because... Δεν είμαι σκιώδης Αντικαθιστώ τον κύριο Όλο Σμιτ που είναι στο Σουρινάμ, που είναι ωραίο μέρος να είναι κανείς, αλλά ήμουν περίεργος. Περίμενα να ακούσω τις εξηγήσεις του συναδέλφου Μπαλτασάρε για να δούμε τι θα γίνει στα τελωνία. Ο κύριος Όλε Σμιτ μου ζήτησε να παρουσιάσω κάποιες παρατηρήσεις του. Ε, είναι ευγνώμων γενικά Θεωρεί ότι είναι σωστή η προσέγγιση του εισηγητή. Για τα τελωνία χρειαζόμαστε περισσότερη ευρωπαϊκή συνεργασία για αποτελεσματική διοίκηση και να αποφύγουμε στρεβλώσεις της εσωτερική αγοράς για το εξελισσόμενο έργο, για το ενωσιακό, την Ενωσιακή Τελωνιακή Ένωση, θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στα συστήματα επικοινωνίας πληροφορίας, και να έχουμε τυποποιημένες διαδικασίες στην Ένωση. Σημαντική και η απλοποίηση για την συμμόρφωση των επιχειρήσεων. Οι οικονομικοί φορείς στην Ένωση και οι επιχειρήσεις που έχουν ε, εξουσιοδοτημένο καθεστώς πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα συγκεντρωποιημένης εκαθάρισης. Δεν πρέπει να περιλαμβάνει χρηματοδότηση ε, μηχανημάτων, ε, μηχανημάτων σάρωσης. Αυτά είναι στο Χέρκυλες. Τώρα δεν είναι εποχή για δαπάνες. Και ο Όλε θέλει να δώσει προτεραιότητα στην ε, πληροφόρηση, ε, επικοινωνία. Ε, οριζόντια πρέπει να δούμε το πρόβλημα μαζί με, όλους, με όλα τα τελωνία. Αυτό θα πρέπει να ε, σε αυτό θα δοθεί προτεραιότητα. Ευχαριστούμε όλους. Αυτά είχα να πω για τον όλες. Η Κομισιόν, πώ θέλει να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Τάσκαλο. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Μπαλτασάρε για την έκθεσή του. Θα θέλαμε να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις για τις διάφορες τροπολογίες που προτείνετε. Καταρχάς, για τις ε, τροπολογίες θα τις ομαδοποιήσω ένα κεφάλαια, δεν θα τις δω μία προς μία, γιατί τελειώς θα καθυστερήσουμε. Um, for all the financial για όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει ένα σχεδιασμό σε τρεις ομάδες, σε γενικούς στόχους, συγκεκριμένους στόχους και επιχειρησιακούς στόχους. Εμείς ε, για το, τα τελωνία του 2020 κάνουμε το ίδιο αυτό τον καταμερισμό και θα θέλαμε να διατηρήσουμε αυτά τα τρία επίπεδα γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ καλύτερη αξιολόγηση των προγραμμάτων και να είναι και συγκρίσιμη με τις υπόλοιπες αξιολογήσεις. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο ανέφερε και σε προηγούμενη συνεδρίαση, στην αρχική έκθεση του κυρίου Μπαλτασάρε, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υποστηρίζει την χρηματοδότηση εξοπλισμού για το πρόγραμμα. Ο προπολογισμό του προγράμματο και το πρόγραμμα αυτό κάθε αυτό δεν έχει σχεδιαστεί για τη χρηματοδότηση εξοπλισμού και θεωρούμε ότι κάποια κράτη-μέλη που ζητούν χρηματοδότηση για τον εξοπλισμό έχουν τρόπο να χρηματοδοτηθούν γι' αυτό. Ένα άλλο στοιχείο αφορά τη συμμετοχή τρίτων χωρών και την εξωτερική διάσταση. Για τις τροπολογίες αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων είναι πολύτιμη για τα προγράμματα. Καταρχά, η συμμετοχή τους είναι περιορισμένη. Είναι περιορισμένη μόνο σε κοινέ δράσεις και όχι σε όλες τις δραστηριότητες. Αυτό αναφέρεται ρητός. Και επίσης, η συμμετοχή προϋποθέτει ότι θα γίνεται κάθε φορά που είναι απαραίτητη, ε, είναι υποέλεγχο, αλλά είναι πάντα ε, πολύ χρήσιμη δεδομένου και του προϋπολογισμού. Και τέλος ένα μικρό σχόλιο για τον ε, προϋπολογισμό που προτείνεται. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό δεν συνάδει με την ευελιξία του προγράμματος, όπως ε, είπαμε και στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριος Μπαλτασάρε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. στην ουσία νομίζω ότι συμφωνούμε. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μάντερς ε, που έλαβε το λόγο εκ μέρους του κυρίου Σμιτ. Εγώ συμφωνώ με τις τροπολογίες του κυρίου Σμιτ, όλες και εν μέρη και με τις ε, τροπολογίες του κυρίου Κοφεράτη. Έχω κάποιες αμφιβολίες στην τροπολογία του κυρίου Κοφεράτη που ζητά να χρηματοδοτηθούν και εξοπλισμός πληροφορικής. Ε, με αυτό τον προϋπολογισμό για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όσον αφορά τώρα τον προϋπολογισμό, θεωρήσαμε ότι καλό θα ήταν να κάνουμε κάποιες ενδείξεις για κάποια ποσά, διότι θεωρούμε ότι μιας κάποιας μορφής κατανομή των πόρων με βάση τις προτεραιότητες ε, που εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να γίνονται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. σε γενικέ γραμμές λοιπόν είναι θετική η στάση μου. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό και με την κυρία Λεγκρίπ για, ε, για το πώ θα οργανώσουμε το διατακτικό που αλλάζει λίγο με τις προτάσεις της, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε συμπεριλάβει τις προτεραιότητες στους συγκεκριμένου στόχους και θεωρώ ότι και αυτό ε, οφείλεται ε, σε μια αίσθηση που θέλουμε να έχουμε ότι εξετάζουμε συνολικά την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, να επιβεβαιώσουμε λοιπόν ε, την ψηφοφορία της 18ης Δεκεμβρίου. Ε, μπορείτε να μεταφέρετε το, το μήνυμα στους απόντες, δηλαδή να λάβουμε υπόψη του συμβασμούς και ε, ψηφοφορία και κλεισμένων των θυρών 18 Δεκεμβρίου. Θα τελειώσουμε τώρα. Ευχαριστώ τους λίγους βουλευτές που βρίσκονται εδώ. Ευχαριστώ και τους άλλους που δεν ήταν εκεί, κυρίως τους χιώδης ηγητές και ευχαριστώ ε, όλους εσάς, την Επιτροπή και για μία φορά τους διερμηνείς, οι οποίοι μπορούν να φύγουν λίγο νωρίτερα. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνετε.